welcome to the second session of the... Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη συνεδρία μας για σήμερα. Θα... Ξεκινήσουμε με μία ενημέρωση σχετικά με την θαυμάσια δουλειά που κάνει η ναυτική μας δύναμη στη Μεσόγειο. Έχουμε την Εούνα Φορμέντ και το διοικητή επικαιρήσεων τον υπονάβαρχο Ενρίκο Κρεντεντίνο, τον οποίο ευχαριστώ για την παρουσία του. Έχει ξανάρθει εδώ στο Κοινοβούλιο ο υπονάβαρχος για τις επιχειρήσει Σοφία και είχατε και την ευκαιρία να τον συναντήσετε στο αρχηγείο της επιχείρησης στην Ρώμη το 16. Όπως ξέρετε, η Σοφία αποτελεί μια επιχείρηση κατά της καταπολέμης, ε, ε, κατά, κατά της διακίνησης ατόμων στην Μεσόγειο. Είναι ένα μικρό κομμάτι της συνολικής προσπάθειας σε σχέση με, την, ε, με το σύνολο της δράσης της Ένωσης και σε άλλους τομείς, ανθρωπιστική βοήθεια, ανάπτυξη, δικαιοσύνη κτλ. Έχω μια στρατηγική αναθεώρηση της επιχείρησης που ξεκίνησε το καλοκαίρι και χωρί μέλη αναμένεται να συμφωνήσουν σε πέντε εβδομάδε σε σχέση με τρει επιλογέ που έχουν ενώπιον του. Καταρχά, η διεύρυνση τη εντολή. Δεύτερον, η διατήρησή τη υπό την τωρινή εντολή με κάποιε προσαρμογέ. Ή τρίτον, το κλείσιμο τη επιχείρηση αυτή. Σήμερα δεν έχουμε ακόμα συμφωνία και η επιχείρηση αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια όπως η ασταθής πολιτική κατάσταση στη Λιβύη που αποτρέπει τις φάσεις 2, β και 3 όπως επίσης τις διαδικασίες εκφόρτωσης αυτών των ατόμων που διασώζονται στην θάλασσα. Υπάρχουν επίσης και συνεχόμενα οικονομικά προβλήματα χρηματοδότησης και κάποιες από αυτές λοιπόν είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Οπότε θα ήθελα, λοιπόν, να να μας ε, δώσετε την άποψή σας σε σχέση με αυτές τις ε, δυσκολίες που αντιμετωπίζετε. Και επειδή γίνονται συζητήσεις μεταξύ των χωρών μελών στο Συμβούλιο για αυτή την επιχείρηση, θα θέλαμε να ακούσουμε και τα επιτεύγματα του Σοφία και τις υπόλοιπες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε. Επίσης θα θέλαμε να ακούσουμε και τις προσδοκίες σας σε σχέση με το μέλλον των επιχειρήσεων αυτών. Υπονάβαρχη, λοιπόν, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι στην Επιτροπή σας. Το 15 είχα ξανάρθει νομίζω. 15-16. Δεκέμβρη 15 τελικά. Είχε μόλις ξεκινήσει η επιχείρησή μας. Τώρα βρισκόμαστε στο τέταρτο έτος επιχείρησης και όπως ξέρετε η εντολή θα εκπνεύσει στο τέλος του τρέχοντος έτους. Και η στρατηγική θεωρήση αναπόκειται στις χώρες μέλη και αναμένουμε την πολιτική απόφαση για την επέκταση της επιχείρησης. Από ό,τι βλέπω υπάρχει βούληση από τις χώρες μέλη για την επέκταση των επιχειρήσεων μέχρι τον Ιούνιο του 20. και έχουμε σχεδόν καταλήξει. Εκριμή παραμένουν τα θέματα της αναδιανομής και της άφηξης στους λιμένες. αποφάσισα πρέπει να ληφθούν στο υψηλότερο το πολιτικό επίπεδο. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν κάποιες συναντήσεις σχετικά με αυτά στο Συμβούλιο και έχουμε τρει μήνε μπροστά μα μέχρι να λάβουμε τελικέ αποφάσει. Θα δώσω κάποια ενημέρωση σε σχέση με την επιχείρηση και τα επιτεύγματά τη και την μελλοντική εξέλιξη, πιθανή μελλοντική εξέλιξη τη επιχείρηση Σοφία, η οποία αποτελεί πήμα τη ευρύτερη προσπάθεια Ένωση για την αντιμετώπιση τη μετανάστευση και στην, ε, συμβάση στην προσπάθεια σταθεροποίηση τη Λιβύης. Η μετανάστευση αντανακλάται σε όλα τα μέτρα που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετανάστευση και την σταθεροποίηση της Λιβύης. Είναι πολύ πολυσχεδής λοιπόν επιχείρηση και θα σας δείξω στη συνέχεια ότι έχουμε καλές διασυνδέσεις με πολλούς διεθνείς οργανισμούς και άλλες υπηρεσίες και όργανα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. το 15 είχαμε αυτό το μοντέλο επιχείρησης και καθήκοντα τα οποία όμως διευρύνθηκαν εντωμεταξύ μετά από την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για το εμπάρκο στη Λιβύη. Παρακολουθούμε μαζί με την ακτοφυλακή της Λιβύης τις ακτές και βοηθάμε τους διεθνείς οργανισμούς και τις αρχές επιβολής αρχής σε σχέση με θέματα διακίνησης σε συνδυασμό πάντοτε με τις λιβικές αρχές. Αλλά θα αναφερθώ σε αυτό αργότερα. Τώρα η κύρια μας εντολή αφορά την κεντρική Μεσόγειο. Δηλαδή την επικράτεια της Λιβύης από τα σύνορα από την Τινησία μέχρι τα σύνορα με την Αίγυπτο. Δηλαδή στο επίκεντρο της κεντρικής Μεσογείου. Συνεργαζόμαστε με διαφορούς φορείς της περιοχής για την θαλάσσια ασφάλεια. Κάπως επικαλυπτόμαστε με την θέμιδα την επιχείρηση δηλαδή της Frontex στην κεντρική Μεσόγειο. Έχουμε το Sea Guardian, άλλη μια επιχείρηση, δηλαδή η ναυτική επιχείρηση που καλύπτει ολόκληρη τη Μεσόγειο και συνεργαζόμαστε με τους ανθρώπου εκεί. Έχουμε επίσης και ανεξάρτητους φορείς και ΜΚΟ που, με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Οπότε έχουμε, όπως βλέπετε, ένα έτσι ευρύ συντονισμό. Τώρα για το κύριο έργο μας. Καταρχάς, εργαζόμαστε ώστε να εξουδετερώσουμε το φαινόμενο της διακίνησης στα διεθνή ύδατα το Phase 2α, όπως λέμε. Έχουμε 51 σκάφη που χρησιμοποιούνται από διακινητές, τα οποία προσπαθούμε να εξετρώσουμε βεβαίω κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και από τότε που ήμασταν ενεργοί είχαν πολλές απώλειες οι διακινητές, λεκούς πόρους, σκάφη, κινητήρες κλπ. Έχουμε επίσης 251 διακινητές ή ύποπτους διακινητές που βρίσκονται στα χέρια των λιβικών αρχών και τώρα έχουμε 45.000 άτομα με τα οποία έχουμε, τα οποία έχουμε διασώσει λιγότερο από το 10% βέβαια του συνόλου που έχουν διασωθεί στην περιοχή. Αυτά είναι τα αποτελέσματά μας. Σήμερα ξέρουν οι διακινητές ότι είμαστε παρόντες και προσπαθούν να μας αποφύγουν εκτός, να πάνε δηλαδή εκτός διεθνών υδάτων της Λιβύης. Ξέρετε ότι η επιχείρησή μας προβλέπε τέσσερις, τέσσερις φάσεις. Εκτός υδάτων, εντός υδάτων συνεργασία με τους Λίβιους και τις Λιβικές Αρχές. Οπότε εδώ αυτό προϋποθέτει πρόσκληση από την Λιβική κυβέρνηση, η οποία πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή ώστε να προσκαλέσει διεθνείς οργανισμού να εργαστούν στην επικρατεία της. Και επίσης θα πρέπει να έχουμε ένα νέο ψήφισμα του ΙΕ, του Συμβουλίου Ασφαλεία, το οποίο θα μα επιτρέπει να πάμε εκεί. Όπω ε, λέγαμε, Πρόεδρε, λόγω τη κατάσταση τη ασφάλεια στη Λιβύη, οι συνθήκες πρόσκλησης μας στη Λιβύη δεν υπάρχουν ακόμα. Εν μεταξύ, στα διεθνή ύδατα προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να φέρουμε σπέρα στην επιχείρησή μας. Για τις μεταναστευτικές δροές. Το 2017 είδαμε ότι οι περισσότεροι μετανάστες που πάνε στην Κεντρική Μεσόγειο προσπαθούν να πάνε στην Ιταλία και από εκεί στην Ευρώπη. Έχουμε την Ανατολική, το Ανατολικό και Δυτικό διάδρομο, αλλά περισσότεροι περνάνε από, το, από την Κεντρική Μεσόγειο. Θα δείτε και του αριθμούς εδώ στα, στις διαφάνειες που έχουμε. Το 2018 άλλαξε η κατάσταση πλήρως. Τώρα δηλαδή ο πρώτος διάδρομος είναι ο δυτικός διάδρομος. 50% των μεταναστών περνάνε από το Μαρόκο στην Ισπανία. 21% παίρνουν τον κεντρικό διάδρομο, κεντρική Μεσόγειος και οι υπόλοιποι την ανατολική, το ανατολικό διάδρομο. Είδαμε μια μείωση 85% των μεταναστών που πηγαίνουν από την ε, Λιβύη στην η Ιταλία σημαντικό, εντυπωσιακό αριθμό αυτό μείωση. Στο κεντρικό λοιπόν διάδρομο είδαμε αύξηση αυτών που πηγαίνουν από την Τινσία στην Ιταλία, αλλά είναι διαφορετική αυτή η μετανάστευση. Είναι περισσότεροι την ίση, οι οποίοι προσπαθούν να φτάσουν στην Ιταλία χωρίς να τους εντοπίσουν. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε. Και θα δείτε ότι η αύξηση της ροής ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2017 και από τότε, όπως είπα, είδαμε ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων που πηγαίνουν από τη Λιβύη στην Ιταλία και βεβαίως είδαμε και μεγάλη αύξηση των θυμάτων στη θάλασσα που πνίγονται. Τώρα υπάρχουν διάφοροι λόγοι για, το, για τους οποίους γίνεται αυτό. Ένας είναι η συνεργασία που άρχισε να φέρνει αποτελέσματα στις χώρες προελεύσης και στη Λιβύη. Υπάρχουν επίσης πολλές δημερείς πρωτοβουλίες μεταξύ, χωρομελών ή με, μεταξύ μερικών χωρομελών και της Λιβύης, μεταξύ αυτών βεβαίως και η Ιταλία. Και το κυριότερο και πιο σημαντικό είναι η εκπαίδευση της ακτοφυλακής και του ναυτικού της Λιβύης μαζί με την αύξηση της ικανότητας και τα σκάφη από το Μάη πέρσι ολοκληρώσαμε την πρώτη φάση εκπαίδευσης και από τον Ιούλιο του 2017 η ακτοφυλακή του ναυτικού άρχισαν να είναι πιο ενεργά στην διάσωση και καταπολέμηση εγκληματικών δραστηριοτήτων και διάσωση ζώων στην Κεντρική Μεσόγειο. Εδώ θα δείτε την συμβολή του ναυτικού και της ακτοφυλακής της επιχειρήσεις διάσωσης και θα δείτε στο πρώτο τέταρτο του 17 είχα ένα συγκεκριμένο σχετικά χαμηλό ποσοστό των επιχειρήσεων το οποίο αυξήθηκε τον Απρίλη αλλά απογειώθηκε το καλοκαίρι βέβαια οπότε στο τέλος του 17 είχαμε 30% επιχειρήσεων, 40% στο πρώτο εξάμεινο και τον Ιούλιο σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων διάσωσης είχαν γίνει από τις ε, λευκές αρχές στην ακτοφυλακή. Μετά βέβαια τον Αύγουστο είχαμε μια έλλειψη καυσίμων και το Σεπτέμβρη στο δικό του τομέα ευθύνη, οι λιβικέ αρχέ και η εκτοφυλακή κάνει το σύνολο των επιχειρήσεων αναζήτηση και διάσωση. Και αυτό το γνωρίζει η διεθνή κοινότητα. Σήμερα λοιπόν η Λιβική Ακτοφυλακή εργάζεται υπό δύσκολε συνθήκε και αναφέρομαι βέβαια στην επίσημη Λιβική Ακτοφυλακή, αυτή που εκπαιδεύουμε, αυτή που ε, είναι υπό τον στρατικό Σεράζη και βλέπουμε ότι γενικά προσπαθούμε να ενισχύσουμε το δυναμικό των λιβικών αρχών. Έχουμε και το εμπάργο ταυτόχρονα το οποίο έχει ένα αντίκτυπο, μια επίπτωση αποτρεπτική κατά το οποίο αναγνώρισε και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και έχουμε κατασχέσει όπλα δύο φορές αλλά επειδή ακριβώς είμαστε πολύ ενεργοί και ορατοί στην κεντρική Μεσόγειο είμαστε παρόντες και μας βλέπουν όλα τα σκάφη που έρχονται από την περιοχή. Έχουμε επαφή με τους διάφορους εταίρους μας και του για την παρουσία μας και τους πληροφορούμε για τις επιθεωρήσεις, τους ελέγχους, ώστε να μην ε, αλωνίζουν ελεύθερα οι διακινητές. Είχαμε και κινητικότητα εντός λιβικών υδάτων αλλά όπως ξέρετε όμως ε, το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας μας επιτρέπει μόνο να δράσουμε στα διεθνή ύδατα. Και αυτό ακριβώς το λόγο θελήσαμε να εκπαιδεύσουμε και τον ναυτικό και την ακτιοφυλακή Λιβύης ώστε να μπορούν οι ίδιοι να παρεμβαίνουν ε, κατευθείαν για να καταπολεμήσουν τους διακινητές και τους ε, εμπορούς όπλων. Και εμείς αν χρειαστεί παρεμβαίνουμε. Γιατί η μάλλον για το λαθρεμπόριο πετρελαίου. Ξέρετε ότι το πετρέλαιο είναι μια από τι κύριε πηγέ εισόδηματο στην Λιβύη, αλλά το λαθρεμπόριο πετρελαίου σήμερα είναι η προπηγή εισόδων για πολλέ δραστηριότητε και οι Λίβοι χάνουν 750 εκατομμύρια ευρώ ετησίως λόγω λαθρεμπορίου πετρελαίου. Υπάρχει δυνατότητα βέβαια πάντοτε ανταλλαγή πληροφοριών και αλλοενημέρωση με του εταίρου μα και υπάρχει δυνατότητα να έχουμε ένα πιο ενεργό ρόλο ώστε να επιθεωρούμε τα σκάφη που ενδεχομένω συμμετέχουν σε αυτό το λαθρεμπόριο. Αποτελεί λοιπόν πρόβλημα για τους ε, Λίβιου το λαθρεμπόριο πετρελαίου. Έχουμε βέβαια ταυτόχρονα και την αύξηση του, της διακίνησης. Αυτά συμβαδίζουν, λαθρεμπόριο πετρελαίου, διακίνηση ατόμων. Ο πρόεδρος Σεράζη ζήτησε από την υπατή εκπρόσωπο να είμαστε πιο ενεργοί στην καταπολέμηση και του λαθρεμπορίου, αλλά εκτός από τη διακίνηση δηλαδή. Και όντως είπαμε ότι για να επιθεωρήσουμε σκάφη θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχουν ύποπτοι και επειδή είμαστε ο μόνος οργανισμός που είναι παρόντας εκεί μα ζήτησαν ακριβώς να καταρτήσουμε και ένα κατάλογο υπόπτων ε, λαθρεμπόρων πετρελαίου. Αυτά λοιπόν για τη Σοφία που δεν σχετίζεται μόνο με την αλλά και με τον ΟΗΕ επειδή μπορούμε να παράσχουμε πληροφορίες και είμαστε εκεί ακριβώς για να δώσουμε ε, πληροφορίες σε όποιον ενδιαφέρεται. και τα στοιχεία που έχουμε ευχαρίστω τα μοιραζόμαστε και με τον ΟΗΕ αλλά και με τους Λίβιους. Εκπαίδευση. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα της επιχείρησής μας. Έχουμε την άδεια να πάμε στα χωρικά υδάτα της Λιβύης αλλά το θέμα είναι οι ίδιοι να μπορούν να καταπολεμήσουν τι εγκληματικέ δραστηριότητε που λαμβάνουν χώρα εκεί και να κάνουν και τι διασώσει. Ξέρετε ότι οι περισσότεροι που πεθαίνουν στην ε, Κεντρική Μεσόγειο είναι στα λιβικά ύδατα ή πολύ κοντά στα λιβικά ύδατα. όπου εμείς δεν παρεμβαίναμε. Και μέχρι το 2017 δεν είχαν καμιά δυνατότητα, καμιά υποδομή για να κάνουν διασώσεις. Τώρα, μετά την εκπαίδευση, και τα σκάφη που έλαβαν από την Ιταλία μπόρεσαν να κάνουν διασώσεις 30.000 περίπου διασώσεις έκαναν τους τελευταίους 15 μήνες και αυτός είναι ένας από τους χειρότερους λόγους που είδαμε την ε, μείωση όσον αφορά τα θύματα πρόσφατα στην Κεντρική Μεσόγειο για την εκπαίδευση. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι εκπαιδεύουμε του σωστού ανθρώπου, του κατάλληλου ανθρώπου και πρέπει να έχουμε μια αυστηρή δικασία επιλογή. Οι χώρε μέλη μαζί με την ε, Europol, μαζί με την Interpol και τι υπηρεσίε πληροφοριών, τι πολιτικέ αλλά και τι στρατιωτικέ συμβάλλουν σε αυτό ώστε να αποδεχόμαστε τους υποψήφιους αφού γίνει μια διαλογή. Και αυτή η διαλογή χρειάζεται περίπου 45 μέρες αφού λάβουμε τα ονόματα των υποψηφίων. Μετά ξεκινάμε την εκπαίδευση. Μέχρι τώρα έχουμε εκπαιδεύσει 238 από τον Αθηγό και την, αγρο... και την ε, λιμενοφυλακή. Στην Ιταλία θα εκπαιδεύσουμε και άλλους, αλλά και αλλού, Κροατία, Ισπανία κλπ. Και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε εκπαιδεύσει γύρω στους 50 ανθρώπους. Οι μισοί εργάζονται στη θάλασσα, οι άλλοι μισοί περίπου στις ακτές, κυρίως στην περιοχή της Τρίπολης. Και είμαι σε επαφή με τους ηθήνοντες της ακτοφυλακής και του ναυτικού. Συναντιόμαστε συχνά, ανταλλάσσουμε πληροφορίες και υπάρχει εμπιστοσύνη και αλληλεγγύη που βεβαίω χτίσαμε μέσω εκπαίδευσης αυτό νομίζω είναι από τα πιο σημαντικά καθήκοντά μας. Η δημιουργία αυτής της αμοιβές εμπιστοσύνης. Στόχος μας παραμένει το να έχουμε εκπαιδεύσει 500 άτομα μέχρι το τέλος του έτους. Αναμένουμε ονόματα από τις λιβικές αρχές και αν η επιχείρηση επεκταθεί, τότε θα συγχρονίσουμε τη δική μας εκπαίδευση με τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λιβύη και τις δράσεις της Ιταλίας, η οποία, στην οποία ανατέθηκε από την Κομισιόν μέχρι το, 2020 ε, να συγκροτήσει το πρώτο κέντρο διάσωσης. Όλα αυτά βέβαια πάντοτε με, σε συνεργασία με τις λιβικές αρχές κυρίως στην Τρίπολη εποπτεία. Είναι ένα καθήκον που μας ανατέθηκε στα τέλη του περσινού και θα πρέπει να δούμε αν όντως πάμε στη σωστή κατεύθυνση, αν οι Λίβοι τα καταφέρνουν, Κάναμε λοιπόν αυτή την εκπαίδευση κυρίως παρακολουθώντας τους στην θάλασσα και χρησιμοποιώντας εξοπλισμό που έχουμε για να κάνουν στη θάλασσα, στην Τίνιδα, στην Ιταλία αλλά και στην Τρίπολη είχαμε κάποιες συνεδριάσεις και εκεί λάβαμε στοιχεία από τις λιβικές αρχές με τις οποίες ούτως ή άλλως ήμασταν σε στενή επαφή και μιλάμε συχνά. Πάντως οι χώρε μέλη επιτρέπεται να κάνουν καθημερινές επισκέψεις ώστε να σχηματίσουν εικόνα. Εγώ αναμένω και την άδεια για την τοποθέτηση δύο αξιωματικών στη Λιβύη, τρει-τέσσερι μέρε τη εβδομάδα, συγγνώμη, ώστε να έχουμε μια αλφα παρακολούθηση και να δούμε ακριβώ τι γίνεται και τι ανάγκε έχουν οι Λίβοι. Αυτά ω τμήμα τη στρατηγική αναθεώρηση και τη συζήτηση για το μέλλον τη Σοφία. Είμαστε πάντως έτοιμοι να τοποθετήσουμε δύο αξιωματικούς αρχικά στην Τρίπολη και μετά που κριθεί απαραίτητο για τρεις-τέσσερις μέρες τη βδομάδα. Αυτό που είδαμε λοιπόν μέχρι τώρα είναι ότι υπάρχουν διάφοροι που επιχειρούν από την Μιζουράτα και από την Τρίπολη. Έχουμε γύρω στις 12-15 εξόδους την εβδομάδα και διάφορες εξόδους χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα σκάφη ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα σκάφη πάνω στη θάλασσα για συντονισμό. Σήμερα μπορούν να εργαστούν μέχρι και το βόρειο κομμάτι, εδώ πέρα το μπλε που βλέπετε στην διαφάνεια της Λιβύης και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον στην Λιβύη και στη Μιζουράτα θα χρησιμοποιούν τα περιπολικά σκάφη που τους έδωσε η Ιταλία. Θα τους δώσουμε άλλα 12 ως Ιταλία, ώστε οι Λίβοι να έχουν ό,τι υλικό χρειάζεται για να περιπονούν σε μια μεγάλη περιοχή. Επίσης, να σας πω ότι έχουμε δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο με συμφωνίας με τις αρχές, επιβολή, με του νόμου και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλε χώρες και από την Ιταλία και σήμερα προσπαθούμε να συμπληρώσουμε αυτό το μοσαϊκό για να καταλάβουμε ακριβώς τι λείπει από αυτή την εξίσωση. Είχαμε και την ε, προσπάθεια για το awareness στην κεντρική Μεσόγειο. Έχουμε συμφωνίες με τις γενικές διευθύνσεις, τις ταλικές για την καταπολέμηση της μαφίας και της τρομοκρατίας και όλοι μαζί σε συνεργασία συντάξαμε την πρώτη έκθεση που αφορά διακινητές και μας δίνει μια καλή εικόνα για το πώς συνδέονται όλα αυτά και βεβαίως είναι ανοιχτό προς συμμετοχή και στους εταίρους μας συνεργαζόμαστε με την Frontex και την Europol και έχουμε ολοκληρώσει ένα κώδικα μαζί με την Κομισιόν και σήμερα στην Αυαρχίδα η οποία αποτελείται από κόσμο της Frontex και άλλους ε, βλέπουμε λοιπόν ότι μέσω αυτού του προγράμματος που θα διαρκέσει ένα εξάμεινο συνολικά θα κρατήσει το πείραμά μας μέχρι τον Νοέμβρη. Πάντως τα πράγματα πάνε μέχρι τώρα καλά και προχωράνε και πρέπει να συνεργαστούμε. Οπότε η εξωτερική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται να συμβαδίζει μέσω επιχειρήσεων όπως η δική μας. Και πραγματικά υπάρχει ένα εντυπωσιακό δυναμικό για την καταπολέμηση οποιασδήποτε εκκληματικής δραστηριότητας. Και αυτό που κάνουμε μέχρι τώρα καταδεικνύει ότι μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Με τη Frontex, η Europol, ανταλλάσσουμε πληροφορίες και αυτό μας επιτρέπει ας πούμε να επιθεωρήσουμε τα σκάφη στην ανοιχτή θάλασσα γιατί για να το κάνουμε αυτό, για να κάνουμε τις επιθεωρήσεις, πρέπει να είμαστε πεπισμένοι ότι υπάρχουν, υπάρχει εμπλοκή αυτών των σκαφών σε εγκληματικέ δραστηριότητε. Έχουν, έχουμε πληροφορίες από τη Frontex και μετά εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Παρέχουμε όμως ε, αντίστροφα και εμείς πληροφορίες στη Europol και την Frontex, ας πούμε, όταν ένα σκάφος φτάσει κοντά στα ύδατα μιας χώρας μέλους, τότε αν υπάρχουν υποψί, ε, υποψίες μπορούμε να επιβαστούμε και να κάνουμε επιθεωρήσεις. Γι' αυτό συζητάμε και για την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Συλλέγουμε πληροφορίε, αλλά και λαμβάνουμε πληροφορίε, βέβαια από την Frontex μέσω των καναλιών που υπάρχουν ώστε να έχουμε μια καλή εικόνα για το τι συμβαίνει και να συμβαδίζουν όλα αυτά με τις αντίστοιχες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτή είναι η προσθέμενη αξία που σας έλεγα προηγουμένως. Είναι λοιπόν σημαντικό να συνεχίσουμε το πρόγραμμα αυτό γιατί περιλαμβάνει μια εσωτερική και μια εξωτερική διάσταση. Τώρα για την Κεντρική Μεσόγειο έχουμε αυτή την ε, εξάμεινη συνάντηση η οποία διεξάγεται σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για θέματα ασφάλειας και διάσωσης στην Μεσόγειο. Φέτος τον Ιούνιο στη Ρώμη είχαμε 242 συμμετέχοντες από πολλές χώρες και πολλούς διεθνείς οργανισμούς. Μέναν μαζί δύο μέρες, είχαμε έξι ομάδες εργασίας που ασχολήθηκαν με διάφορα θέματα η μια αξία όμω το να μείνουμε όλοι μαζί, να παραμένουμε ενωμένοι, να συζητάμε, να δράσουμε πληροφορίε κλπ. Γιατί όλε οι ΜΚΟ που δουλεύουν στην ε, Μεσόγειο είναι πολύ σημαντικέ και θα ξανασυνδεθούμε στα τέλη του Νοεμβρίου Ρώμη. Και πάλι σημαντικό είναι η κοινότητα του εμπορικού ναυτικού. Κάποιες λοιπόν ομοσπονδίες και οργανώσεις ναυτιλιακές εμπλέκονται εδώ και θέλουμε να κάνουμε κάποια διάσκεψη μαζί τους. Έγινε ήδη μία στο Λονδίνο και η δεύτερη ήταν τον περασμένο μήνα στο Αμβούργο με τη Γερμανική Ομοσπονδία. Πάντως θα πρέπει όλοι να συνεργαστούμε, όλοι εμπλεκόμενοι δηλαδή στην Κεντρική Μεσόγειο. Συμπράσματα και θα σταματήσω να απαντήσω στα ερωτήματα σας αν έχετε. Άτυπη μετανάστευση, μάλλον παράτυπη μετανάστευση από τη Λιβύη έχει δραστικά μειωθεί 86% σε με πέρσι. Τώρα κατά πόσο αυτό είναι βιώσιμο δεν το ξέρουμε, κανείς δεν μπορεί να πει. Αυτό που ξέρουμε ότι στη Λιβύη σήμερα υπάρχουν 600.000 άτομα και έχουμε να κάνουμε με κόσμο που έχει χάσει τα πάντα λόγω πολέμου σε μια χώρα η Λιβύη που παραμένει πλούσια. Αναμένουν λοιπόν την σταθεροποίηση της χώρας και να επανέλθουν στην κανονική του ζωή. Αλλά 300.000 άτομα είναι μετανάστες, είναι έτοιμοι να μετακινηθούν, οπότε θα μπορούσαν και πάλι να βγουν στη θάλασσα και να πάνε στην Ευρώπη μέσω Ιταλίας. Ή θα, θα μπορούσαν να προσπαθήσουν εναλλακτικέ οδούς όπως Μαρόκο Ισπανία. Τι θα γίνει στο μέλλον δεν ξέρουμε, αλλά θέλουμε να παραμείνουμε παρόντες εκεί και είναι γι' αυτό το λόγο σημαντικό να διατηρήσουμε την σοφία, η επιχείρηση δηλαδή τη Ένωσης στη Κεντρική Μεσόγειο, που παρουσιάζει στρατηγικό ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το capacity building ένα σημείο κλειδί, εκπαίδευση της ακτοφυλακής και του ναυτικού, ώστε να ενστερνιστούν τις προσπάθειες αυτές οι Λιβύοι. Όπως είπε και ο πρόεδρος της Λιβύης. Είναι σημαντικό λοιπόν να διευρύνουμε την εκπαίδευση και στις υπόλοιπες δυνάμεις ασφαλείας της χώρας. Σήμερα, όπως ξέρετε, είναι μια πολύ ασταθής χώρα η Λιβύη, κάτι σαν τη Σομαλία. Πρέπει λοιπόν να σταθεροποιήσουμε τη Λιβύη, διαφορετικά δεν θα μπορούμε να κάνουμε κάτι σοβαρό. Για το εμπάργκο όπλων. Έχουμε αποτρέψει τη διακίνηση των όπλων στο εσωτερικό της Λιβύης και για το λαθρεμπόριο έχουμε καταλήξει πια σε μια κατανόηση του φαινομένου αλλά χωρίς τους Λίβιους τους ίδιους δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και αυτό ακριβώς θα πρέπει να έχουμε και εμείς και έναν πιο ενεργό ρόλο εδώ. Και όπως είπα πριν, συνδέουμε την εσωτερική με την εξωτερική διάσταση στις επιχειρήσεις μας. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό και είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτά είχα να πω. Είμαι στη θέση σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα ε, ενημερωτική και μερικές φορές ε, θετική παρουσίαση ε, της δουλειάς που κάνετε εδώ και πολύ καιρό και τη διαφορά που κάνει για τις ζωές των ανθρώπων.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 από καρδιάς ε, τον ομιλητή για τις ε, πληροφορίες που μοιράστηκε μαζί μας, ε, που είναι πάρα πολύ επίκαιρες και πρόκειται επίσης για πληροφορίες πολύ υψηλής ποιότητας. Το να μειώσουμε τη μετανάστευση σε αυτό το τμήμα του κόσμου σημαίνει ότι μειώνεται και ο απολογισμός σε ανθρώπινες ζωές και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να σας κάνω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δορυφορικές εικόνες, ας πούμε το Κοπέρνικους, ε, για άμεση αναγνώριση, να δείτε το, το, το μέγεθος του φαινομένου, να χρησιμοποιείτε για παράδειγμα δεδομένα που έχει στη διάθεσή της η Frontex και επίσης τα δισεκατομμύρια που χάνονται στο λαθρεμπόριο πετρελαίου. Έχετε ιδέα των διαδρομών των ε, λαθρεμπόρων αυτών και πού πηγαίνει όλο αυτό το πετρέλαιο. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Τέζα. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίζω τον υπονάβαρχο ο οποίος μας κάνει περήφανος στην θέση του ως υπεύθυνος του Σοφία. Το λέω αυτό ω Ευρωβουλευτής, ως Ιταλός και ίσω στην Ιταλία έχω κατανοήσει πλήρως την σημασία του ρόλου του. Έχουν γίνει γιγαντία βήματα χάρη ακριβώς στην επιχείρηση Σοφία. Ίσως λοιπόν Πρόεδρε θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην επικοινωνία μας προς τα έξω για να καταστήσουμε κατανοητό ποιο ήταν ο ρόλο τη Ευρώπη μέσω τη επιχείρηση Σοφία. Όχι μόνο στη διάσωση ανθρωπίνων ζώων κάτι το οποίο είναι προφανές πέρα από τις κουβέντες μας και τις πολιτικές συζητήσεις αλλά επειδή τελικά μέσω των σκαφών που εσείς καθοδηγείτε έχουμε σώσει πολλές ζωές Αυτό δεν είναι και τόσο γνωστό γιατί θεωρεί ο κόσμος προς τα έξω ότι έχει άλλη είδους δράση η Σοφία. Αλλά κυρίως έχουμε να κάνουμε διάσωση ανθρωπίνων ζωών και αποτροπή των διακινητών και αντιμετώπιση βεβαίω και του λαθρεμπορίου πετρελαίου. Και κυρίως το γεγονός ότι πήγατε στη Λιβύη για να εκπαιδεύσετε αυτούς που σήμερα από ό,τι είδαμε στο γράφημα από το Σεπτέμβρη το 90% των ατόμων που σώθηκαν, σώθηκαν ακριβώς από την ακτοφυλακή της Λιβύης με τη δική σας βοήθεια. Αλλά και από την Ιταλία, έτσι να το πούμε ξεκάθαρα, από την Ιταλία που παρήχε υλικό, σκάφη κλπ. Αλλά λοιπόν πραγματικά που στην Ιταλία δεν είναι πλήρως κατανοητή και γνωστή η δουλειά που κάνετε. Αυτά που κάνουμε συνολικά ως Ευρώπη στην Μεσόγειο δηλαδή. Να κλείσω το εξή. Όταν μας λέτε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι πιο ενεργή, τι εννοείτε. Βεβαίως πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την επιχείρηση. γιατί 400.000 άτομα που είναι εκεί και θέλουν να φύγουν θα αποτελούσαν ένα μελλοντικό πρόβλημα για μας. Οπότε όταν λέτε η Ευρώπη πρέπει να είναι πιο ενεργή τι εννοείτε, απτά συγκεκριμένα, τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω για να πετύχουμε αυτά που λέτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους δύο συναδέλφους ε, και θα ήθελα και εγώ ε, ως πρόεδρος ε, να κάνω κάποιες ερωτήσεις, να σχολιάσω και κάποια εξ όσων αναφέρατε. Να συνεχίσω αυτό που είπατε, αλλά μόνο, όχι μόνο για την Ιταλία. Νομίζω το ευρύτερο ζήτημα της επικοινωνίας σε σχέση με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας επειδή έρχονται και εκλογές ε, το 2019 στους πολίτες μας καλύτερα τι έχουμε επιτύχει. Καταλαβαίνω ότι είναι περισσότερο δική μας ευθύνη και όχι δικός και ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε καλύτερα πώς θα διαφημίσουμε την επιτυχία στον τομέα αυτόν θα ήταν νομίζω πάρα πολύ χρήσιμο. Κάτι ακόμη που θα ήθελα να σχολιάσω. Μιλήσατε ότι χρειάζεται μία ε, απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, εν είδη follow-up Χαίρομαι που άκουσα για την επιτυχία του πιλωτικού προγράμματος ε, και ε, για, την ανταλλαγή απόψεων που υπήρξε και με την ευρωπαϊκή πλευρά. Υπάρχει περαιτέρω δράση που θα πρέπει να καλυφθεί και στο πλαίσιο του επόμενου πι. Μήπως πρέπει κάπως να θεσμοθετήσουμε, για να το πω έτσι, τα ε, επόμενα βήματα και σε σχέση με αυτό. Και κάτι ακόμη το οποίο ε, θέσατε επίσης για τη συνεργασία με τους μη κυβερνητικού οργανισμούς. Προφανώς υπήρξε πολλή κάλυψη των συγκεκριμένων οργανισμών ε, στην Μεσόγειο και θα με ενδιαφέρε να μου πείτε πώς συνεργάζεστε μαζί τους. Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο περισσότερα για αυτά. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε ακόμη πολλά περισσότερα να ρωτήσουμε σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε αυτές τις ερωτήσεις. Θα απαντήσω στα Ιταλικά αν δεν σας πειράζει. Εποφελούμε της προηγούμενη παρέμβασης. Για να πω ότι για μένα είναι τιμή μεγάλη που ηγούμε αυτές τις ευρωπαϊκές αποστολές. Για τους δορυφόρους να σας πω ότι χρησιμοποιούμε ευρέως τους δορυφόρους, τους ευρωπαϊκούς, σε συνεργασία με τη Frontex. Η Frontex αποτελεί την πρώτη οντότητα, τον πρώτο οργανισμό με τον, οποίο είχαμε συμφωνία. Έχουμε αυτή την αδελφή επιχείρηση, όπως τη λέμε, που είχαμε με τη Frontex από την αρχή και κάναμε εξοικονομήσεις και εναλμονήσεις στα πλαίσια του προπολογισμού που έχουμε. ιδιαίτερα για τη χρήση των δορυφορικών εικόνων. Το πρόβλημα με τι δορυφορικέ εικόνε είναι ότι είναι πολύ σημαντικέ από στρατηγική σκοπιά, όμω για άμεση δράση, τακτική δηλαδή η δράση, η αποτελεσματικότητα είναι χαμηλή, επειδή δεν υπάρχει χρόνο για λήψη, εξέταση κλπ. Γι' αυτό ακριβώ είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τα drones. Εμείς είχαμε κάποια από αυτά τα μηχανήματα μας έδωσε η Ιταλία που αποδείχθηκαν τελικά κρίσιμα. Γιατί όταν πετά το drone, εγώ άμεσα λαμβάνω πληροφορίες βιντεοσκοπημένες στο κέντρο ελέγχου και μπορώ να καθοδηγήσω τις δράσεις. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Τα drones δεν χρηματοδοτούνται από κοινωτικά κονδύλια σήμερα χρηματοδοτήθηκαν για μια πειραματική περίοδο η οποία έχει ολοκληρωθεί. Είχαμε και μια έκθεση προς τις χώρες μέλη σχετικά. Οι χώρες μέλη βέβαια αποδέχτηκαν την έκθεση σκεπτόμενες ότι θα μπορούσε να υπάρξει συνέχιση της ε, χρηματοδότησης. Τα αεροπλάνα είναι πολύ χρήσιμα αλλά εξίσου χρήσιμα είναι και τα drones, τα οποία ακριβώς εντοπίζουν πρώτα τα σκάφη και μας ε, στέλνει τις εικόνες. Το αεροπλάνο μπορεί να ε, βρίσκεται στον αέρα μόνο 2-3 ώρες. Το drone αντίθετα 10-12 ώρες. Και η πτήση στα όρια των διεθνών υδάτων επικίνδυνη περιοχή, έτσι, γιατί δεν ξέρει κανεί τι γίνεται. Αν καταρρύψουν ένα ντρόν, εντάξει, δεν έγινε τίποτα, δεν έχουμε πιλότου, μόνο οικονομική απώλεια. Με τα αεροπλάνα το αντίθετο. Έχουμε λοιπόν ευελιξία με τα ντρόν που δεν μα παρέχει κανένα άλλο μέσο. Γι' αυτό ακριβώ θα πρέπει να πείσουμε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το μηχανισμό Αθηνά, δηλαδή κοινωτικά κονδύλια, ακριβώ για να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα. Και αυτό το συζητάμε ακόμα στι στρατηγικέ μα συζητήσει. Τι μου είπατε. Α, να μιλήσω πιο αργά για τους διερμηνείς. Εντάξει. Τα χρησιμοποιούμε λοιπόν όλα αυτά. Τώρα. Στρατηγική επικοινωνία. Ήθελα και εγώ να το σχολιάσω αυτό. Ε, δεν γίνεται σε δικό μας επίπεδο, αλλά σε υψηλότερο επίπεδο. Βρυξέλλες και χώρες μέλη. Εγώ το κάνω επειδή είχα κάνει και δραστηριότητες εξωτερικών σχέσεων είχα εκπροσωπεύσει την Ένωση στην Αντιζαμπέπα, τον ΟΗΕ επίσης και λοιπά και λοιπά. Και στο εξωτερικό προσκλήθηκα την περσμένη εβδομάδα στην Ουόσιγκτον από τον επικεφαλής άμυνας της, τον ΙΠΑ, με 80 επικεφαλής άμυνας από άλλες χώρες και του μίλησα για την επιχείρηση Σοφία. Σοφία που είναι μια επιχείρηση που γνωρίζουν στην Ουάσιγκτον και αλλού. Δεν θέλω όμω να κάνω κάτι τέτοιο ως στρατηγική επικοινωνία. Πρέπει να γίνει σε πιο ψηλό επίπεδο. Εμείς αν κάνουμε μόνο διασώσει, θα είχαμε βάλει τα σκάφη μα μπροστά στη Λιβύη και θα είχαμε σώσει τον κόσμο. Αλλά δεν είχαμε εντολή να κάνουμε κάτι τέτοιο. Είχαμε εντολή να χρησιμοποιήσουμε τα σκάφη μα για να καταπολεμήσουμε για κινητέ, όχι για να σώσουμε τον κόσμο. Είναι δύσκολο λοιπόν να σώσει τόσο, πολλο, τόσο πολύ κόσμο, 45.000 κόσμο, μια μεγάλη χώρα. Πάντως, καταπολεμήσαμε τους διακινητές εξωτερώνοντας τα σκάφη που χρησιμοποιούσαν τα οποία δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιήσουν δημιουργώντας τους απώλειες είχαν ας πούμε μεγάλα καΐκια που χρησιμοποιούσαν τα οποία ήταν τελείως ανασφαλή και ήταν αυτά που οδήγησαν στα μεγάλα ατυχήματα στα, μεγάλα ναυάγια, Λαμπεντούσα και αλλού Καταπολεμούμε επίσης και τους εμπορούς και ελαθρεμπόρους όπλων. Τους ελαθρεμπόρους όπλων. Για το λαθρεμπόριο πετρελαίου. Σύμφωνα με την εντολή μου, αυτό που μπορώ να κάνω μόνο είναι το να συλλέξω πληροφορίες. Και πώς το κάνουμε αυτό. Βλέπουμε, ας πούμε, αν το τάνκερ έχει τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει, αν έχει τη σωστή σημαία ευκαιρία, αν έχει αλλάξει νεολόγια, αν έχει αλλάξει εφοπλιστή. Έχουν το ολοκληρωμένο σύστημα εντοπισμού, μάλλον ταυτοποίηση. τα τάνκερ τα οποία παρέχουν πληροφορίε όταν βρίσκονται εμπλό. μετά από κάποια χωρητικότητα, κάποιο εκτοπισμό, εκτόπισμα και πάνω. Αν δούμε, ας πούμε, ότι σβήνουν αυτό το σύστημα ε, ταυτοποίησης και μετά το βρίσκουμε μπροστά μας σε μια απομακρυσμένη ακτή της Λιβύης αυτό το τάνκερ, ε, τότε καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Στη Μάλτα σε διεθνή ύδατα υπάρχει μια τοποθεσία που έχουμε και νόμες αλλά και παράνομες δραστηριότητες. Θα δείτε στη φωτογραφία εδώ ότι γίνεται μετάγγιση πετρελαίου από ένα τάνκερ σε άλλο. Και εδώ ακριβώς το ντρόν μας επέτρεψε να εντοπίσουμε αυτή την συναλλαγή που ήταν λαθρεμπόριο. Και μετά βέβαια το πετρέλαιο αυτό διαχείριται παντού στην Ευρώπη, πάει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και μετά και μέσω Σουέζ στην, ενδικό Ινδικό ωκεανό. Αλλά κυρίως πάει από τη Λιβύη στη Μάλτα και μετά σε ευρωπαϊκές χώρες. Και γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό να έχουμε ένα πιο ενεργό ρόλο, δηλαδή να μπορέσουμε να επιθεωρούμε τα τάνκερ γιατί έχουμε ένα κατάλογο το οποίο καταρτίζουμε με υπόπτη που παραδίδουμε στον ΟΗ, αλλά με τι επιθεωρίε επιτόπου μπορεί να έχουμε τη βεβαιότητα τέλο πάντων ότι πράγματι αυτό το τάνκερ συμμετέχει, εμπλέκεται σε αυτό, την, σε αυτό το λαθρεμπόριο. ώστε μετά να αναλάβουν οι αρμόδιες αρχές άλλων χωρών. Θα μπορούσαμε επίσης να σταματήσουμε ή να κατασχέσουμε και τα τάνκερ, αλλά έστω και μία επιθεώρηση αρκεί για να διαπιστώσουμε κατά πόσο εμπλέκονται στο λαθρεμπόριο αυτά τα τάνκερ, να ενημερώσουμε μετά τις χώρες του νεολογίου και μετά να προβούμε στις απαραίτητες συλλήψεις. Για την ακτοφυλακή της Λιβύης από τότε που κάνει διασώσεις η ακτοφυλακή η Λιβική είδαμε αυτή τη μείωση του 80% για δύο λόγους. Καταρχάς, επειδή αυτό είχε τεράστιες επιπτώσεις στους διακινητές, ας πούμε, πριν να παρεμβούν οι Λίβοι, οι διακινητές, δεχόταν μια προκαταβολή από τους μετανάστες. Δηλαδή, πριν την αχώρηση πήραν από το ταξίδι τους. Τώρα που ξέρουν ότι πολλοί μετανάστες θα γυρίσουν στη Λιβύη, οι διακινητές θα πληρωθούν το σύνολο μόνο όταν είναι βέβαιοι οι μετανάστες ότι θα φτάσουν στη χώρα προορισμού. Αυτό έχει αντίκτυπο και στους ίδιου του μετανάστες γιατί σήμερα οι μετανάστες ξέρουν ότι πάρα πολλοί θα διασωθούν από την ακτοφυλακή και θα επαναοδηγηθούν στην Λιβύη. Οπότε είναι σημαντικό για αυτούς να αναζητήσουν εναλλακτικέ οδούς από τη Λιβύη. Γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδεύσουμε τους Λίβιους από την κυβέρνηση Σεράζη και να παρακολουθούν, να υποπτεύουν και να διασφαλίσουμε τέλο πάντων ότι δουλεύουν σωστά και ότι τηρούν τους διεθνείς νόμους και το κοινοτικό δίκαιο. Να σου πω επίσης ότι η εταίρη μας στην εκπαίδευση είναι η υπατερμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, η Frontex, η Έχουμε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, έχουμε θέματα φύλου και ε, κάναμε και μια εκπαίδευση ε, στους Λίβιους για θέματα φύλου, οι οποίοι θα γίνουν μετά μετεκπαιδευτές ακριβώς για θέματα φύλου. Να σκεφτείτε ότι στην ακτοφυλακή στο ναυτικό της Λιβύης δεν υπάρχουν γυναίκες. Ο στρατός ναι έχει γυναίκες, αλλά όχι το ναυτικό και ακτοφυλακή. Από τότε λοιπόν που ξεκινήσαμε την εκπαίδευση για το θέμα φύλου, άρχισαν να προσλαμβάνουν και γυναικείο προσωπικό, το οποίο είναι βασικό. Πολύ σημαντικό. Τώρα, για τον ΟΗΕ. Για να πάει κανείς στα χωρικά έντατα της Λιβύης, χρειάζεται ή απαιτεί τέλο πάντων ένα ψήφισμα του ΟΗΕ. Όμως για να βγει αυτό το ψήφισμα του ΟΗΕ, χρειάζεται συνένεση προφανώς ή συγκατάθεση της λιβικής κυβέρνησης. Και κάποιες χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν θα συμφωνήσουν ποτέ Όλα αυτά συνδέονται. Εμεί λοιπόν μπορούμε να πάμε στη Λιβύη κατά πάσα πιθανότητα μετά τις εκλογές στη Λιβύη. Να δούμε λοιπόν αν αυτές οι εκλογές θα οδηγήσουν σε πιο σταθερή κυβέρνηση, αλλά μέχρι να συμβεί αυτό, εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στην Λιβύη, στα διεθνή ύδατα, και να πενθυμίσω, όπως έλεγα πριν, ότι η Σοφία αποτελεί μια επιχείρηση θαλάσσιας ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε η παρουσία μας δεν αποσκοπεί μόνο στην καταπολέμηση του, του λαθρεμπορίου των διακίνητρων και διάσωση ε, ζώων, αλλά ξέρουμε ακριβώς εμείς τι γίνεται ως πολεμικό ναυτικό και μπορούμε να προσφέρουμε πληροφορίες στις χώρες μέλη σε σχέση πούμε, με τρομοκράτες που φτάνουν στα στις θάλασσες αυτές. Ή να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση οποιαδήποτε ε, ε, κίνηση γίνεται εμπορικής φύσης σε αυτή την περιοχή. Ευχαριστώ. Thank you very Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρώτησα και για το follow-up του πιλωτικού προγράμματος. Μήπως θα θέλατε να πείτε και κάτι σε σχέση με αυτό. Για το πιλωτικό του Νεύρη θα υποβάλουμε τα αποτελέσματα με τους διευθυντές Europol Front, Frontex κλπ. Είμαι όμως παπισμένος ότι αφού τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά και ορατά και το δυναμικό είναι τεράστιο, αυτό θα κάνουμε. Δηλαδή να έχουμε στρατιωτικές επιχειρήσεις με πολιτική διάσταση επίσης σε συνεργασία με τι αρχέ επιβολής του νόμου, με τι οποίε είναι ξεκάθαρο πρέπει να συνεργαστούμε. Δεν μπορεί καθένα να δουλεύει μόνο του, χωριστά οι στρατιωτικοί, χωριστά οι πολίτε. Η συνεργασία μεταξύ των δύο είναι κάτι το καθοριστικό για το μέλλον και αυτό ακριβώ έχει ξεκινήσει με την επιχείρηση Σοφία. Thank you very much. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που είπατε ότι θα έπρεπε να σας συγχαρωτήσει ποιος είναι ο ρόλος των γυναικών σε τέτοιες καταστάσεις. Ε, ε, ε, ήρθα σε κάποια μηχανία, αλλά εν πάση περιπτώσει ευχαριστώ πολύ που το είπατε αυτό και που είπατε ότι υπάρχει συνέχιση αυτής της τάσης της πρόσληψης στην UNAFOR για την Μεσόγειο επειδή είναι ιδιαίτερε οι συνθήκες. Επίσης είναι πάρα πολύ χρήσιμο να έχουμε όλη αυτή την ενημέρωση που μα ε, κάνατε σήμερα όσον αφορά την επιτυχία, την εξέλιξη της δουλειάς που κάνετε, που περάσατε από τη μετανάστευση στο θέμα του λαθρεμπορίου, πετρελαίου και ε, εργάζεστε υπό διάφορους ε, τρόπους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε ευγνώμονες για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής μας και της δουλειάς που κάνετε. Ευχαριστούμε και πάλι θερμότατα για την παρουσία σας ε, και βεβαίως θα είμαστε σε επαφή. So, colleagues, briefly uh, Απλώς να σας ενημερώσω σύντομα ε, ότι 4 η ώρα πρέπει να αρχίσουμε με το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξής μας. Ε, περιμένουμε τους συναδέλφους να, έρθουμε, να έρθουν, τους συναδέλφους που θα παρουσιάσουν το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει λοιπόν μία σύντομη διακοπή, αλλά παρακαλώ να είστε πίσω εγκαίρως. Ευχαριστώ. Good afternoon. And, uh, again... Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο, στη δεύτερη συνεδρία της απογευματινής μας, το δεύτερο τμήμα της απογευματινής μας συνεδρίας που θα εστιαστεί στην δράση για τις νάρκες και την ολοκληρωμένη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη δράση για τις νάρκες. Πρόκειται για ανταλλαγή απόψεων με τον Φρανκ Μόισεν που είναι αρμόδιος για θέματα πολιτικής, συμβατικά όπλα αφοπλισμός, Φωτεινή Αντωνοπούλου, Διευθύντρια Προγράμματος Επικεφαλής της Δράσης για τις Νάρκες, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, Συνταματάρχης Φραντς Επικεφαλής Κοινών Στρατιωτικών Υποθέσεων, Αντιναρκικό Τμήμα στη Δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα από την επιχείρηση Αλτέα και ο Χουάν Κάρλο Ρουάν, που είναι διευθυντής της Μονάδας υποστήριξη τη εφαρμογή της Σύμβασης για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού από το Διεθνές Κέντρο Άρσης Ναρκοπαιδείων για ανθρωπιστικούς σκοπούς της Γενέβης. Και τέλος, Αλέξη, σου σημαντική, είναι η Jane Κόκκινγκ, διευθύνουσα σύμβουλος από τη συμβουλευτική ομάδα και τις νάρκες. Ένας ε, από τους λόγους της ε, σημερινής μας ε, συνεδρίας είναι να προσπαθήσουμε να γνωστοποιήσουμε περισσότερο και να ενισχύσουμε την προσπάθεια αυτή που γίνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είναι ένα ζήτημα συνεχές. Στις 30 ε, Σεπτεμβρίου, πριν από 10 μέρες, ε, τρία παιδιά σκοτώθηκαν και ένα τραυματίστηκε όταν στην Ανατολική Ουκρανία ε, εξεράγει μία ανάρκη αυτό μας, θυμάζει, μας θυμίζει το, την τεράστια πρόκληση, την ανθρωπιστική ε, που ε, αποτελεί, ε, οι, αποτελούν οι νάρκες και άλλοι εκρηκτικοί μηχανισμοί. Οπότε οι συνάδελφοι είναι εδώ για να συζητήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Χαίρομαι που έχουμε μαζί μας ένα πάνελ ε, ε τέτοιων εμπειρογνωμόνων και με πολύ χαρά περιμένω να ακούσω από εσά πώς είναι η κατάσταση γενικότερα στην ε, δράση για τις νάρκες ε, σε σχέση με την εκστρατεία ε, γης χωρίς νάρκες μέχρι το 2030. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε αυτή τη δράση και πώς αυτό συμπληρώνει την ε, δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα στον τομέα αυτό. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μέρσεν, θα πείτε κι εσείς φαντάζομαι μερικά πράγματα γι' αυτό εδώ το έγγραφο που σας δείχνω αυτή τη στιγμή, που είναι υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δράση για τις νάρκες σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχει στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα ισπανικά, εδώ μπροστά, στο μπροστινά έδρανα, ε, στην αίθουσά μας, αν οι συνάδελφοι θέλουν να ε, τα πάρουν. Αυτό είναι εν μέρει ένα τμήμα, ε, μια εισαγωγή στην παρουσίασή σας. Έχετε το λόγο κυρία Μαϊσέν; Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας που που κάλεσε την ΕΕ, Είναι πάρα πολύ σημαντική ανταλλαγή απόψεων για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τις νάρκες. Δυστυχώς ο ειδικό απεσταλμένος για τη μη ε, διάδοση, ο κύριος ε, Βιλίτσα, είναι στη Νέα Υόρκη για, την πρώτη, για τη συνεδρίαση της πρώτης επιτροπής του ΟΗΕ. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μακρά ιστορία υποστήριξης της δράσης για τις νάρκες, κάτι εποφελές για όλες τις χώρες ε, και τις περιφέρειες του κόσμου. Ε, είναι ο δεύτερος ε, δωρητής, όπως είπε και η Πρόεδρος. Τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση για την απαγόρευση των ναρκών και έχουν υποστηρίξει την οικουμενικοποίηση της σύμβασης αυτής η υποστήριξη ε, καλύπτει ολόκληρη, ολόκληρο το φάσμα της ε, δράσης ε, για τις νάρκες, η εκπαίδευση για τους κινδύνους, η απελευθέρωση της γης και η αποναρκοθέτηση, η καταστροφή των αποθηκών, η ενίσχυση των θυμάτων, μεταξύ άλλων. Οι νάρκες βρίσκονται στο σταυροδρόμι ε, πολλών ε, διαφορετικών ε, τομέων και διαστάσεων. Υπάρχει η διάσταση της ασφάλειας, της ανθρωπιστικής βοήθειας, της σταθερότητας σε τομείς μετά ε, από ε, πολεμικές ε, συγκρούσεις, όταν δηλαδή κάποιες περιοχές, οποίες βέβαια υπάρχουν οι αλλά το ξέρει ο κόσμος και δεν πηγαίνει σε αυτές τις περιοχές και δεν, είναι, δεν απειλείται η ζωή κανενός, όμως υπάρχουν κάποιες κοινωνικές και κοινωνικές παράμετροι που επηρεάζουν κατά άλλο τρόπο αυτές τις περιοχές. Για παράδειγμα, δεν μπορούν να τις εκμεταλλευτούν γεωργικά. Υπάρχει ένας κοινωνικο οικονομικο αντίκτυπος πολύ σημαντικός λοιπόν. Υπάρχει και η πτυχή της ανάπτυξης. Υπάρχει επίσης ε, το θέμα των, ε, των θυμάτων, άνθρωποι που αποκτούν αναπηρίες και χρειάζονται ειδική ε, υποστήριξη για το υπόλοιπο της ζωής τους και υπάρχει μάλιστα και συνθήκη που καθιστά υποχρεωτική την εκαθάριση από νάρκες ε, ακόμη και αν δεν υπάρχουν ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές πτυχές που να συνδέονται με ένα ναρκοπαίδιο. Από το 2001 στο 2008 η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ένα συγκεκριμένο συγκεκριμένο οικονομικό μέσο που αφορούσε τη δράση για τις νάρκες, όμως στο πλαίσιο των διαφόρων ε, ε, διαστάσεων και πτυχών που σας έδειξα προηγουμένως, το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να συμπεριληφθεί η διάσταση της ε, δράσης για τις νάρκες σε, διάφορες θεματικές, σε διάφορα θεματικά και γεωγραφικά μέσα. Αυτό σημαίνει αποκέντρωση, αύξηση της ευελιξίας και επίσης αυξήθηκε και ο συνολικός προπολογισμό που αφιερώθηκε σε αυτό το σκοπό, όμως η αρνητική πλευρά είναι ότι χάνεται ε, το κατά ε, ε, η, το, το, η αίσθηση του πόσο, εφικτού είναι τα, πόσο εφικτά είναι τα πράγματα, όπως επίσης και η καθοδήγηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα υπήρξε και ένα ερώτημα από τους συναδέλφους σας πέρσι, για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υποστηρίζει την δράση για τις νάρκες. Μα είναι ο δεύτερος υποστηρικτής παγκοσμίω. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικό δωρητή, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα εφικτότητας. Ε, αυτό λοιπόν ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει πιο αισθητή η δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, να την επικοινωνήσουμε καλύτερα μέσω όλων αυτών των ευρωπαϊκών μέσων και μέσω όλων αυτών που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2001 ε, ε, και μετά. Αυτή η προσπάθεια έχει εντατικοποιηθεί μετά το 2016. Βλέπετε εδώ την υποστήριξη ε, σε 33 χώρες σε όλο τον κόσμο σε όλες τις υπηρούς σχεδόν ε, για 300 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Αυτή η υποστήριξη έλαβε χώρα μετά με διάφορους τρόπους, ε, με, με προσαρμοσμένους τρόπους ανάλογα με τις ιδιωτερότητες των διαφόρων ενδιαφερομένων χωρών και μιλάω όταν λέω για, ε, για επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εννοώ τα κράτη-μέλη, εννοώ τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και τα κράτη-μέλη είναι επίσης σημαντικά. Ε, εδώ βλέπετε επίσης τους βασικούς αποδέκτες ε, της χρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσης για τις νάρκες. Καλύπτει τις χώρες ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κροατία, η οποία είναι μεταξύ των 10 πιο πληγισών χωρών στον κόσμο, έχει λάβει 84 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή... 58% ε, του ποσού. Υπάρχουν βέβαια διαφορετικά μέσα χρηματοδότησης που προέρχονται και από άλλα, ε, από άλλα μέσα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, οι Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειών και Ανάπτυξης επίσης συμμετέχουν με έναν προπολογισμό ειδικό, ο οποίο όμω είναι ξεχωριστό από τον, ε, ε, από τον ε, προπολογισμό υποστήριξης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε εδώ τους 50 πιο σημαντικού εταίρους. Βλέπω εδώ τη σύμβαση της ε, ΟΤΑΒΑΣ ε, που εκπροσωπείται σήμερα ε, και άλλος ένας εταίρος εκπροσωπείται εδώ σήμερα. Κατά τη γνώμη μας η δράση αυτή είναι αποτελεσματική με μεγάλη υποστήριξη, με ευρύτερη υποστήριξη, αποτελεσματική υποστήριξη. Δηλαδή και από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών σε συνεργασία με τους δωρητές αλλά και με την ε, ε, κοινωνία των πολιτών. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο των ε, πράξεών μας, των δράσεών μας. Γνωρίζετε όμως ότι η εθνική κυριότητα χρειάζεται τεχνογνωσία, χρειάζεται υποδομή και οι δωρητές έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν στην ανάπτυξη των χώρων, ε, των χωρών μενάρκες στην ανάπτυξη των χωρών μενάρκες τη δική του ικανότητα να αντιμετωπίσουν επίση το πρόβλημα. Βλέπετε ότι από το 2012 μέχρι το 2016 ε, η η τα μεγαλύτερα, τα πιο σημαντικά προγράμματα είναι το UNDP και το UNMAS όσον αφορά τη χρηματοδότηση δράσης ναρκών. Ε, προφανώς θα, ε, ε, ε, δουλέψει κανείς σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, των κρατών, συγγνώμη, με Ε, όμως, σε Πολλέ περιπτώσεις όταν πρόκειται για μετασυγκρουσιακέ περιπτώσεις έχουμε ε, το UN ενώ σε ε, χώρες όπου δεν υπήρχε τόσο πολύ αυτό το, ε, αυτά τα κλασικά προβλήματα των μετασυγκρουσιακών περιόδων είναι το UNDP. Βλέπετε εδώ το χρηματοδοτικό μέσο που πιο πολύ συνεισφέρει στη σταθερότητα είναι το ICSP ε, βάσει του άρθρου 3, το ICSP υποστηρίζει συχνά τη δράση για που καλύπτει την υποστήριξη των χωρών ε, ακόμη και στην πρόληψη των ε, συγκρούσεων και έχει και μια αναφορά στη δράση των ναρκών, κατά των ναρκών σε πολλές περιπτώσεις ε, είναι τμήμα της ε, αναπτυξιακής βοήθειας. Ε, για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει μια χρηματοδότηση μέσω του DCI ή του Ταμείου Ανάπτυξης από τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ ή στο πλαίσιο μιας προταξιακής βοήθειας από τη Γενική Διεύθυνση ΝΙΕΡ ανάλογα με την χώρα για την οποία πρόκειται. Υπάρχουν επίσης και κάποια κατασπέσεις κατά πιστεύματα όπως το Σαχέλ, το Μαντάτ που χρησιμοποιούνται για τέτοιου είδους ε, χρηματοδότηση στην περίπτωση ανθρωπιστικών, ε, ανθρωπιστικών ε, καταστάσεων είναι περισσότερο η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ. Υπάρχουν και κάποια εσωτερικά μέσα, στην περίπτωση της Κροατίας για παράδειγμα, και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πάρει την απόφαση της οικουμενικοποίησης της σύμβασης της Οτάβας, ε, Η ομάδα υποστήριξης για την εφαρμογή της σύμβασης προσπαθεί να ε, ε, βοηθήσει ε, την ομάδα του Συμβουλίου που ασχολείται με αυτό. Θα το αναφέρει φαντάζομαι ο συνάδελφος. Αλλά νομίζω σημαντικό είναι να πούμε ότι οι αποστολές στρατιωτικές και μη στρατιωτικές πολιτικές μπορούν να βοηθήσουν στις δράσεις αυτές. Τώρα, συχνά λαμβάνουμε ερωτήματα από τους εταίρους μας, ε, πώς να προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τη δράση για τις νάρκες. Να πάτε στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην χώρα για την οποία πρόκειται. Ε, σε τρίτες χώρες οι αντιπροσωπείες έχουν πολύ σημαντικές για τον προγραμματισμό και την ε, κατανομή της χρηματοδότησης ε, γιατί ξέρουν πολύ καλά τη χώρα και μπορούν να έρθουν σε επαφή με το πιο κατάλληλο μέσο και είναι πάρα πολύ καλό ότι είναι εδώ το ότι έχουμε έναν συνάδελφο από την επιχείρηση Αλθέα να μας παρουσιάσει την εμπειρία ε, μπορείτε λοιπόν να μάθετε με ποιον πρέπει να έρθετε σε επαφή ε, μέσω της αντιπροσωπείας. Μερικά πράγματα τώρα για την πορεία από εδώ και στο εξής. Ε, ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται αυτή τη στιγμή επί του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, δηλαδή του προϋπολογισμού 2021 έως 2027 και το ζήτημα είναι ποια θα είναι η θέση της δράσης ε, για τις νάρκες στο πλαίσιο αυτό. Ο ρόλος ε, θα συμπεριληφθεί σε διάφορες θεματικές ενότητες ή θα είναι κάτι διαφορετικό. Κάτι ακόμη, να έχουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, κάποιους προσανατολισμούς. Έχουμε ήδη, αλλά να πρέπει να αναθεωρηθούν, να επικαιροποιηθούν. Ίσως με την ε, αναθεώρηση της ε, σύμβασης της ΟΤΑΒΑ του χρόνου, που θα γίνει ε, του χρόνου στο Όσλο, με το νέο σχέδιο δράσης για τα επόμενα πέντε έτη. Αυτό νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να ενημερώσουμε και την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΝΑΡΚΕΣ. Και επίσης υπάρχει και το θέμα του 2025 την προηγούμενη, ε, στην προηγούμενη προσπάθεια αναθεώρησης στο Μαπούτο, τα κράτη-μέλη δεσμεύθηκαν σε μια φιλοδοξία για έναν κόσμο χωρίς νάρκες μέχρι το 2025. Ε, και μάλιστα η υποχρέωση αυτή είναι αρκετά ισχυρή. Διάβασα η Νότια Κορέα και η Βόρειος Κορέα συμφώνησαν να αποναρκοθετήσουν στο όριο, ε, στο σύνορο μεταξύ τους. Που είναι ένα ε, ναρκοπαίδιο το οποίο είναι από τα γνωστότερα στον κόσμο. Αν εξαφανιστεί αυτό το ναρκοπέδιο, αυτό είναι μία ακόμη όθηση για την πλήρη ε, εξουδετερώση των ναρκοπαιδίων παντού. Επίσης, ε, αυτοσχέδιες ε, χώρε, ε, συγγνώμη, νάρκες κατά προσωπικού στο, στο Ιράκ, στη Λιβύη. Ε, αυτές οι αυτοσχέδιες νάρκες είναι ένα φαινόμενο αύξων. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κανείς κατασκευασμένες βιομηχανικώς νάρκες. Αυτό δείχνει αυτό το φαινόμενο του αυτοσχεδιασμού. Γι' αυτό οι ενδιαφερόμενοι προσπαθούν ε, να τα ε, κατασκευάσουν μόνοι τους, γιατί είναι αδύνατο νομίμως να βρεθεί αυτό το προϊόν. Η σύμφαση της Οτάβας σημαίνει πολυμερισμός ε, στην καλύτερη, στην του εκδήλωση, γιατί από 163 ε, μέλη, συμβαλόμενα μέλη, έχει απαγορευτεί, έχουν απαγορευτεί κάποια όπλα, Υπάρχουν όμως κάποιες προκλήσεις ακόμη, γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτό το ορόσημο ε, πολυμερισμού θα εξακολουθεί να ε, ισχύει και στην περίπτωση της δράσης για τις νάρκες, γιατί οι νάρκες είναι κάτι το οποίο είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να επιληθεί. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μην μας διαφεύγει και έτσι κλείνω και την παρουσίασή μου. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που τονίσατε μία ακόμη φορά την πολύ σημαντική δουλειά ε, που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και όλα αυτά που πρέπει να εξετάσουμε από εδώ και στο εξή. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στο δεύτερο, στη δεύτερη ομιλήτριά μας, συγγνώμη, στον ομιλητή μας ε, που αναφέρθηκε ήδη, το συνταγματάρχη Φραντ Λόρσινγκ, ο οποίος έχει μια πραγματική εμπειρία της επιχείρησης Αλθέα στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ε, θα ε, δώσω αρχικά το λόγο στην ε, συνάδελφο Φωτεινή Αντωνοπούλου διότι μοιράσαμε την παρουσίασή μας σε δύο μέρη. προετοιμάσαμε την παρουσίαση αυτή από κοινού με κάλεσαν σήμερα με τον συνταγματάρχη Λέσνινγκ για να σας παρουσιάσω το πώς η ε, αντιπροσωπεία της, Ευρωπαϊκής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, Βοσνία Ερζεγοβίνη αντιμετωπίζουν το ε, πρόβλημα, της, το ζήτημα της δράσεως των ναρκών χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Δράσης από το 2016. Οι πρώτες δύο διαφάνειες ίσως να είναι μικρές και δύσκολες να διαβαστούν από μακριά. Αρχικά έχουμε το ε, πώς την δημιουργία ικανοτήτων ε, στην Βοσνία Ζεργοβίνη όπου χρησιμοποιούμε δύο πολιτικές από τη μία θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές ε, περιβάλλον και το επιτυγχάνουμε αυτό χρησιμοποιώντας τα προενταξιακά ε, ταμεία, είπα, ε, υποστηρίζοντας τις τοπικές αρχές ούτως ώστε να βελτιώσουν τις δυνατότητές τους και ε, σε δράσεις σε καθαρισμού των ναρκών. Ε, επίσης χρησιμοποιούμε τον μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα και ειρήνη που αναφέρθηκε νωρίτερα καθώς επίσης ε, και την U4 Althea. Ο δεύτερος στόχος είναι να, να βοηθήσουμε τις ικανότητες της χώρας για μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και το χρησιμοποιούμε αυτό ε, με, ε, χρησιμοποιώντας ε, ποσά για τον καθαρισμό ναρκών, την εκπαίδευση, την βοήθεια θυμάτων. Όλα αυτά έχουν μια άμεση θετική συνέπεια στην οικονομική ανάπτυξη, όμως η εκαθάριση ναρκών ταυτόχρονα σημαίνει και την δημιουργία προγραμμάτων ε, υποδομών, ενισχύει την ε, συνοριακή ασφάλεια και επίσης υπάρχουν και ποσοτικά ε, στοιχεία που το επιδεικνύουν, όμως δεν ετοιμάσαμε έναν ολόκληρο κατάλογο των επιτευμάτων μας. Η πρόεδρος ζητάει να σταλούν αργότερα. Αυτό το οποίο θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας εδώ στην είναι ότι η Επιτροπή επισκέφθηκε νωρίτερα την ε, ε, Βοσνία Ερζεγοβίνη και είχε τη δυνατότητα ε, να συζητήσει με εμπειρογνώμονες, με εκπροσωπήσεις θυμάτων, με οργανώσεις που κάνουν τους καθαρισμούς και είδαν επίσης τις δυνατότητες που έχει ε, μία μονάδα που είναι υπεύθυνη για την ε, αποναρκωθέτηση. Το η U4 έχει επίσης ε, μία χρόνια παρουσία στην χώρα, όμως η εκαθάριση αρκών ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια με στόχο να παράσχει υποστήριξη όσον αφορά την εκαθάριση και ταυτόχρονα να ε, παράσχει και την αναγκαία εκπαίδευση, μόρφωση. Ε, επίσης υπήρξε ένα πιλωτικό ε, πρόγραμμα το οποίο έδειξε ότι η ε, προσέγγιση απελευθέρωσης γεών είναι ιδανική για την χώρα και μπορεί να εφαρμοστεί και σε μεγαλύτερο βαθμό. Όσοι δεν γνωρίζετε είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος ο οποίος εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες. Μενάρκες το υποστηρίζει ο ΙΕ καθώς επίσης και πολλές ε, άλλες, ε, άλλες διεθνείς οργανώσεις, όπως και το Διεθνές Κέντρο Άρσης Ναρκοπαιδίων για Ανθρωπιστικούς Σκοπούς της ε, Γενέβης. Υποστηρίζονται τέτοια προγράμματα, καθότι στην Βοσνία Ζεγοβίνη δεν υπάρχουν πολλά τέτοια. Ένα από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής προγραμμάτων από το 2012 και έπειτα ήταν το γεγονός ότι οι εταίροι μας έπρεπε να καθαρίσουν περιοχές ε, όπου εν τέλει δεν υπήρχαν καθόλου νάρκες ε, ή οι βασικές πληροφορίες ήταν πέρα ως πέρα λάθος, με αποτέλεσμα να σπαταληθούν ε, πόροι Η υποχρέωσή μας ε, λοιπόν να παράσχουμε βοήθεια με αποτελεσματικότητα και ταυτόχρονα να δείξουμε στους Ευρωπαίους φορολογούμενους ότι η βοήθειά μας, ε, ότι η βοήθειά μας ε, προς τις χώρες πραγματικά φέρει αποτελέσματα. Μας έκανε να σκεφτούμε έξω από τα συνηθισμένα και κάναμε μια συνεργασία με την U4 για να ταυτοποιήσουμε τα προβλήματα και να βρούμε από κοινού λύσεις και καθώς επίσης με τη βοήθεια των εθνικών εταίρων. Όμως, ε, καθώς ε, ε, επεκτείναμε τα χρονοδιαγράμματα, συνεργαζόμασταν, προσπαθούσαμε να βρούμε αποτελεσματικές λύσεις από άποψη ε, κόστους. Κάθε μέρα στην Βοσνία Ζεγοβίνη κόσμος τραυματίζεται ή και πεθαίνει. Έτσι είναι η κατάσταση λοιπόν όταν ένα τρακτέρ ε, μπει σε μια χωροθετημένη περιοχή ή που μπορεί να μην είναι χωροθετημένη. Αυτό ήταν ένα ατύχημα πέρσι τον Σεπτέμβριο. Ε, δύο νεκροί. Τα τελευταία εννέα χρόνια που συμπίπτουν ε, και με την ε, στρατηγική για τις νάρκες που υιοθέτησε το 2009 η χώρα υπήρξαν 132 θύματα, 53 εκ των οποίων ε, σκοτώθηκαν. Οι περισσότερες, οι πιο επηρεασμένες κοινότητες είναι αυτές οι οποίες ε, βρίσκονται κοντά σε δάση, έχουν χωράφια τα οποία δεν μπορούν να καλλιεργήσουν. Ε, πολλές οικογένειες, πολλές περιοχές παραμένουν ανασφαλείς. Πολλοί τυχαίνει, πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν στα δάση παρά τις ε, προειδοποιήσεις. 20 χρόνια μετά τη λήξη του πολέμου στο μέσο της Ευρώπης η Βοσνία Ερζεγοβίνη ε, θεωρείται ακόμα μία από τις ε, χώρες με τις περισσότερες νάρκες στον πλανήτη. Οι περισσότερες περιοχές, νάρκες βρίσκονται στις ζώνες ε, διαχωρισμού Βοσνία, Αρζεγοβίνη στα σύνορα ε, με την Κροατία καθώς επίσης και στην ε, Δημοκρατία της Σέρβσκα υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα ενώ υπάρχουν και περιοχές από που έχουν αφαιρεθεί νάρκες και έχουν μεταφερθεί σε αγνωστές περιοχές από το 2018 προσπαθούν να ανταποκριθούν στις ε, προσπάθειες καθαρισμού. Τα τελευταία χρόνια μονάχα το 50% των ε, στόχων έχουν καθαριστεί και παρόλο που οι δωρεές συνεχίζουν να καταφθάνουν ε, με τον κλασικό ρυθμό, η μονάδα απομάκρυνση ναρκών που βρίσκεται υπό την εντολή των ενόπλων δυνάμεων έχει συνεισφέρει ιδιαίτερος ε, σε αυτό το 50% παρόλο που σίγουρα θα είχε καταφέρει πολλά περισσότερα. Ο ε, συνταγματάρχης Λέσνινγκ τώρα θα σας εξηγήσει για ποιο λόγο ε, το εναπομείνον έργο φαίνεται τόσο δύσκολο ε, και και για, ποιο για λόγο χρησιμοποιήθηκαν ε, χρήματα από το Μηχανισμό Συμβουλής στη Σταθερότητα και Ειρήνη, ούτω ώστε να βοηθηθεί η χώρα. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητά μέλη, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να συνεχίσω και να ε, τονίσω τους ε, βασικούς ε, λόγους που υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Αρχικά βλέπουμε ότι υπάρχει μία ανάγκη καλύτερης ευθυγράμμισης της στρατηγικής με την πραγματικότητα που υπάρχει κατά τόπους, καθώς επίσης και τις υποχρεώσεις και τα χρονοδιαγράμματα. Η Βοσνία έχει αποτύχει να επιτύχει να τον στόχο απομάκρυνση όλων των αρκών, όμως υπάρχουν αδυναμίες μεταξύ της, ε, του συστήματος διαχείρισης ε, ποιότητες ε, και των συστημάτων που υπάρχουν και παρόλο που υπάρχει η δυνατότητα καλού ελέγχου, η συνολική, το συνολικό σύστημα θα πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ. Ορισμένες διαδικασίες από την άλλη ε, συνεχίζουν να μην υπάρχουν ενώ όταν εφαρμόζονται φαίνεται ότι δεν ακολουθούν τα μαθήματα που, του παρελθόντος. Το περιβάλλον θα πρέπει να προσαρμοστεί όπως ε, το διαχειριζόμαστε τώρα. Έχουμε μια, έναν κατάλογο ε, χιλίων στόχων. Είναι εμφανές λοιπόν όταν, ότι όταν έχεις τόσες πολλές προτεραιότητες ε, δυσκολεύει στην επίτευξη των στόχων και στο να υπάρχει μια στοχευμένη προσέγγιση. Θεωρούμε λοιπόν ότι το ε, PHMAC θα πρέπει να βελτιωθεί ιδιαιτέρως, ε, ιδιαιτέρως όσον αφορά την ε, αποστολή πληροφοριών, τις εκθέσεις, πέραν τούτου. Η συνάδελφος ανέφερε ήδη ότι τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν δεν καλύπτουν όλη την Βοσνία με με αποτέλεσμα πολύ συχνά να υπάρχουν ε, λαθασμένες πληροφορίες ε, και πράγμα το οποίο προσθέτει ένα επιπλέον άχθος. Τέλος, ε, η πολύπλοκη διοικητική δομή της χώρας φαίνεται από τα διάφορα κυβερνητικά ε, ιδρύματα και τους παράγοντες οι οποίοι συμμετέχουν ε, στην όλη διαδικασία στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Αυτός ο χάρτης που βλέπετε μπροστά σας σας ε, δείχνει πώς είναι η κατάσταση. Όπως βλέπετε υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι συμμετέχουν στην απομάκρυνση ναρκών. Έχουμε την μονάδα απομάκρυνσης ναρκών, έχουμε ΜΚΟ, έχουμε την κυβέρνηση, έχουμε διμερείς δωρεές και προγράμματα, έχουμε 26 παράγοντες οι οποίοι συμμετέχουν κατά τόπους, όμως ε, δεν έχουμε μια στρατηγική προσέγγιση ε, κατά τόπους. Ε, τώρα πώς συνεισφέρει η EU4 στην όλη προσπάθεια στην Βοσνία Ερζεγοβίνη. Αμέσως μετά το τέλος ε, του πολέμου ξεκίνησε τις δράσεις απομάκρυσης ναρκών ε, και υποστήριξε την Ευρω... τον ΟΗΕ και την ΜΑΚ ε, και υπήρξε μια έντονη συνεργασία στην χώρα καθώς επίσης και με τις εθνικές αρχές. Η κοινότητα απομάκρυνσης ναρκών οργανώθηκε γρήγορα με υποστήριξη από διεθνείς ε, παράγοντες. Υπήρξε μια επιτροπή απομάκρυνσης ε, ε, ναρκών, επίσης υπήρξε ομάδα από τον ΟΗΕ. Στη συνέχεια εφαρμόστηκε μια στρατηγική έγιναν πολλές προσπάθειες και όλα αυτά είχαν την υποστήριξη της EU4 ε, και ε, με αυτόν τον τρόπο μειώθηκε ο ρόλος ε, της U4. Στην αρχή είχαμε 44 άτομα προσωπικό, τώρα είμαστε στα 11. Ο ρόλος λοιπόν προσαρμόστηκε στην κατάσταση. Αυτό το οποίο κάνουμε ακόμα είναι ότι στηρίζουμε την μονάδα απομάκρυνσης ναρκών όμως ε, ταυτόχρονα παρακολουθεί και το έργο της επιθεωρώντας τις δράσεις κατά τόπους, δίνει συμβουλές, ε, μεταφέρει πληροφορίες σε, όλους, σε όλα τα συμμετέχοντα ε, μέρη. Τώρα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Αποστολή παρέχει συμβουλές, δίνει τεχνικές πληροφορίες και αυτά λοιπόν είναι, είναι πράγματα τα οποία θα συνεχίσουμε και όσον αφορά ε, την εφαρμογή των ε, προγραμμάτων τα οποία αναφέρθηκαν ήδη από τη συνάδελφο. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι γνωρίζετε το συγκεκριμένο ε, project, γι' αυτό το λόγο θα αναφέρω τα βασικά στοιχεία στοχεύουμε το πρόγραμμα Find a Job να ε, ταυτοποιήσει ε, περιοχές ε, με νάρκες από διάφορες περιοχές, να μειωθεί ο αριθμός των τοποθεσιών από 8.600, οπότε θα μειωθούν οι προτεραιότητες που έχουμε και θα έχουμε και μία νέα βάση δεδομένων στο πλαίσιο του UNTP και θα έχουμε και ένα νέο σύστημα προτεραιοτήτων. Η EU4 θα συμμετέχει στο Διοικητικό ε, Συμβούλιο, θα λαμβάνει αποφάσεις ε, για όλο αυτό το ε, πρόγραμμα εκπροσωπείται και η αποστολή της, Ευρωπαϊκή, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό και στη συνέχεια θα ενημερώνει την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ούτω ώστε να τους δίνει πληροφορίες για να λαμβάνουν τις αναγκαίες αποφάσεις. Θα θέλαμε να τονίσουμε λοιπόν ότι τα τελευταία τρία χρόνια καταφέραμε με επιτυχία να ενσωματώσουμε ε, τρία διαφορετικά εργαλεία χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο πολύπλοκο τομέα της απομάκρυνσης της ναρκών και ελπίζουμε ότι ε, μπορούμε έτσι να συνεισφέρουμε ούτως ώστε η Βοσνία Ζεγοβίνη να επιτύχει ε, να φτάσει πιο κοντά στους στόχους της συνθήκης της, ΟΤΟ, της ΟΤΑΒΑ και μέχρι το 2025 δεν θα έχει καθόλου νάρκες πλέον. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την επεξήγηση σχετικά με την κατάσταση στη βοσνια Πριν περάσουμε όμως τους τελευταίους ε, δύο ομιλητές, ε, και εξετάσουμε τον ε, γενικότερο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την απομάκρυνση των ε, ναρκών. Ένας συνάδελφος είπε ότι θα πρέπει να φύγει, οπότε Τζέφρι, αν θέλεις να ε, μιλήσεις. Παρακαλώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που έχουμε αυτή την ευκαιρία. Τι ωραία μουσική ήταν στα αυτιά μας αυτά που ακούσαμε από τους τελευταίους ομιλητές. Ε, πραγματικά είμαι περήφανος ε, για το γεγονός. Ε, εγώ ήμουνα την δεκαετία του 90 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα ήμουν πρωτοστάτης στο να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα θύματα των ναρκών και με την αποναρκοθέτηση και νομίζω ότι ήμασταν και πρωτοστάτες στην, στην, στο να γίνει η σύμβαση η πρώτη του 1999. Οπότε πραγματικά έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλη αυτή την ιστορία. μου και εισηγητής ε, για την έκθεση του Κοινοβουλίου το 2011. Ενδεχομένως ε, καλό θα ήταν ε, να γίνει μία ακόμη έκθεση που θα μπορέσει και αυτό να συμπεριληφθεί στο σύστημα. πραγματικά Αυτά που ακούσαμε σήμερα ε, εδώ είναι πράγματα που τα συζητούσαμε και πριν από 21 χρόνια. Τότε είχαμε πει ότι αυτό έπρεπε να είναι ένα πεπερασμένο πρόβλημα. Έχουμε τόσες, τόσους πολλούς πόρους ε, να διαθέσουμε. Μέσα σε 10 χρόνια θα έπρεπε να έχουμε τελειώσει με αυτό το θέμα. Ε, τώρα όμως έχουμε φτάσει το 2018. βλέπουμε τέλος πάντων ότι μάλλον είναι φαίνεται το τέλος αυτής της διαδικασίας επιτέλους στον ορίζοντα. Το ελπίζω, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν πολλά προβλήματα ε, τα οποία τονίσατε. Καταρχάς, ε, στο παρελθόν ήμασταν πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ ε, καλοί ε, στο να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα ε, θεωρούσαμε δηλαδή ότι μια και είμαστε δυτικές δημοκρατίες μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να λύσουμε αυτό το πρόβλημα ειδικά όταν αντίπαλοι μας είναι τρομοκράτες ε, οι οποίοι δεν έχουν κανένα σεβασμό για την ανθρώπινη ζωή το γεγονός ότι είναι επίσης, γεγονός είναι επίσης ότι ένας από τους μεγάλους συνεισφορείς ε, στη δράση για τις νάρκες είναι και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, πρέπει να το πούμε και αυτό. Τώρα, η ανθρωπιστική εκαθάριση των αρκών από ναρκοθέτηση ε, σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει 100% ασφάλεια. Είπατε κι εσείς ότι έχετε εξοδέψει πολύ χρόνο και πόρους ε, σε καθάριση περιοχών όπου δεν υπάρχουν νάρκες, αλλά υπάρχει μια ιδέα ότι υπάρχει απειλή νάρκης. Ε, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γιατί οι τεχνολογίες πάντα προσπαθούν να βρουν αυτήν την μαγική λύση για να μας βοηθήσουν να δούμε πού ακριβώς υπάρχει το πρόβλημα. Αυτό λοιπόν λοιπόν φαίνεται να συνεχίζεται. Επίσης πιστεύαμε ότι πολλές χώρες, εσείς μιλήσατε για τη Βοσνία συγκεκριμένα, ε, δεν έκαναν αρκετά για να βοηθήσουν εκείνοι τους εαυτούς τους και μας αυτό που μας ανησυχούσε τότε είναι τότε γιατί οι ένοπλες δυνάμεις δεν είναι εκπαιδευμένες για δράση ε, κατά των ναρκών ώστε να μπορούν να λάβουν περισσότερη δράση σε αυτό το τομέα. Χαίρομαι που υπάρχει ένα τάγμα από ναρκοθέτηση στη Βοσνία αυτή τη στιγμή Ε, ε, Βέβαια, το στρα... η στρατιωτική αποναρκοθέτηση είναι διαφορετική από την ανθρωπιστική, γιατί είναι το, επίπεδο, το θέμα είναι το επίπεδο του κινδύνου που είναι αποδεκτό. Προφανώ είναι διαφορετικό, αλλά σε μία περίοδο ειρήνη μπορεί να ζητήσει κανεί διαφορετικά πράγματα από το στρατό και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να μην μπορεί να κάνει την ανθρωπιστική αποναρκοθέτηση και άλλωστε αυτοί που την κάνουν οι περισσότεροι είναι πρώην στρατιωτικοί. Άρα, εν πάση περιπτώσει, η καλύτερη στόχη εξειδίκευση είναι πολύ σημαντική. Ε, το είπατε κι εσείς. Ε, πραγματικά με μεγάλη αγωνία θέλω να δω πώς θα γίνει αυτή η καλύτερη στόχευση που λέτε τώρα και σε αυτό το τομέα και σε πολλούς άλλους. Ε, και επίσης υπάρχει το θέμα του συντονισμού των πόρων ε, ιδανικά ενδεχομένω μέσω του ΟΗΕ, μέσω των κέντρων δράσης για τις νάρκες, ανθρώπους που ε, πιέσαμε πριν από πολλά χρόνια και βλέπω με χαρά ότι εξακολουθεί να ε, έχει κάποιο νόημα. Εντάξει, η καταθλιπτική πλευρά είναι ότι ακόμη το συζητούμε και έχουμε φτάσει το 2018, αλλά σημειώνουμε πρόοδο, καλή πρόοδο, και αν ο ορίζοντάς σας είναι το 2025, αν ε, εκπληρωθεί αυτός ο στόχος, τότε πρέπει να ε, στοχεύσουμε καλύτερα ε, τους πόρους μας και πρέπει οι ένοπλες δυνάμεις να αξιοποιηθούν περισσότερο σε ενδιαφερόμενες χώρες για ε, να ξεπεράσουμε το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μήπως μπορείτε να μας πείτε και τους ιστοτόπους σας για περισσότερες πληροφορίες. Ίσως θα μπορούσατε να τις δώσετε στο προσωπικό της Επιτροπής μας, στη Γραμματεία, για να μας τα διαβιβάσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζέφρι. Βλέπουμε Βλέπω ότι χαίρεσαι και είναι λογικό να χαίρεσαι που βλέπεις ε, ότι καρποφόρησαν οι προσπάθειες και οι δικές σου ε, στη Βοσνία Ριζεγοβίνη. Να δώσω τώρα το λόγο στους επόμενους δύο μιλητές και μετά θα επιστρέψω στους συναδέλφους για περισσότερες παρεμβάσεις. Να σας ε, παρουσιάσω τώρα τον κύριο Ρουάν, που είναι διευθυντή της Μονάδας Υποστήριξης εφαρμογή σύμβαση για την Απαγόρευση των Αρκών κατά προσωπικού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα να είμαι εδώ, να σας ενημερώνω και είναι καλό να ξέρω ότι υπήρχαν άνθρωποι, υπάρχουν εδώ άνθρωποι που ήταν εδώ τη δεκαετία του 90 γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό ε, να είναι εδώ μαζί μας αυτοί οι άνθρωποι και στις συζητήσεις αυτές. Ναι, μιλούσαμε για τα ίδια πράγματα νομίζω και πριν ε, από τόσα χρόνια. Ίσως έχουν αλλάξει το, αλλάξει το πώς κάνουμε τα πράγματα πλέον, ε, η επαγγελματική προσέγγιση, αλλά έχετε απόλυτο δίκαιο ότι τα προβλήματα προβλήματα που υπήρχαν τότε εξακολουθούν να υπάρχουν και σήμερα. Χουάν ε, Κάρλο Ρουάν λέγομαι, είμαι διευθυντή τη ομάδα υποστήριξη εφαρμογή τη σύμβαση. Για 11 χρόνια πιο πριν ήμουν ε, ε, στη Ουάσιγκτον και δούλευα σε χώρες της Κεντρικής Αμερικής, στην Ικαράγουα κλπ. Ε, στην σύμβαση της Γενέβας, στο πλαίσιο της Γενέβης, είμαστε σε ένα μικρό κομμάτι της Γενέβης ε, στο, στο ευρύτερο διεθνές τμήμα υποστήριξης της δράσης των αρκών και ε, έχουμε εδώ και κάποια χρόνια αφιερωθεί ε, στην εφαρμογή της, στην υποστήριξη της εφαρμογής σε χώρες όπως το Αφγανιστάν για παράδειγμα όπως γνωρίζετε υπάρχει απειλή σε αυτή τη χώρα εμείς λειτουργούμε με θελοντικές συνεισφορές από πολλά κράτη-μέλη επίσης στηρίζουμε τις ε, συνεδριάσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως, ε, μια ετήσια ανεπίσημη ε, συνεδρίαση και, και αναθεώρηση, διάσκεψη αναθεώρηση της σύμβασης κάθε πέντε χρόνια. Μετά από τη 17η συνεδρίαση των συμβαλωμένων κρατών, η Προεδρία θα αναλυφθεί από την Νορβηγία και θα έχουμε τη διάσκεψη αναθεώρηση την επόμενη χρονιά, κάτι που μας δίνει πολλές ευκαιρίες, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, για να γίνουν σοβαρές αλλαγές, πραγματικές αλλαγές στον τρόπο που θα προχωρήσουμε. Όπως είπε ο Φρανκ, είμαι πάρα πολύ περήφανος ε, γιατί ε, υποστηρίζω την εφαρμογή ενός μιας απόφασης του Συμβουλίου. Ε, αυτή η προσπάθεια οικουμενικοποίησης, ε, καθάρισης των ναρκών, άρσης των ναρκών, αυτό, έχει γίνεται εδώ και τρία χρόνια και μέχρι το 2020 είχαμε πάει στη Βαγδάτη πριν από λίγες εβδομάδες για ενίσχυση των θυμάτων. Στην Καμπάλα πήγαμε επίσης, την επόμενη εβδομάδα θα πάμε στο Σεράγεβο και στις αρχές Νοεμβρίου θα πάμε στη Σενεγάλη για να δούμε πώς είναι η κατάσταση άρσης των αρκών εκεί. Πολλοί από εσά μπορεί να μην ξέρετε από πού προέκυψε η σύμβαση αυτή, αλλά θα ήθελα να τονίσω κάτι τέτοιο, κάτι που θα σας δείξω τώρα και στην οθόνη, ε, δείχνει πολλά για το πού βρισκόμαστε υπήρχαν, ε, αυτό ουσιαστικά ε, προέκυψε από την κατάσταση στην Καμπότζη όταν είδαμε πόσοι πολλοί τραυματισμοί, πόσε ζωές χάνονταν, ακροτηριασμοί από τα πεδία μάχης ε, και λέγαμε μα τι γίνεται, νομίζουμε ότι είμαστε σε περίοδο ειρήνης, όχι πολέμου. Αυτό μας το είπαν οι Human Rights Watch και άλλες συμβουλευτικές ομάδες και ζήτησαν να πιέσουμε για την απαγόρευση των κατά προσωπικού, κάτι το οποίο έγινε το 1997. Αυτή, αυτή η, φωτογραφία λοιπόν δείχνει ο Ζων Κασέ που ήταν ε, ο πρώην ε, προ, πρωθυπουργός του Καναδά Κόφι Ανάν ε, ο Κορνίλιος Ενερούγκα, πρόεδρος του RCRC και η Τζόντι Βίλιαμς που Είχε πάρει τον Νομπέλ Ειρήνης ε, για τη δουλειά με την κοινωνία των πολιτών. Ε, ε, συμμετείχαν σε αυτήν την σύμβαση το 1997 για την απαγόρευση των αρκών κατά προσωπικού. Πήρε όμως πολύ καιρό να συνασπιστούμε γύρω από όλον αυτόν τον αγώνα και είχε μια επιρροή στον τρόπο με τον οποίο κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Εγώ είμαι στη Γενέβη και βλέπω πώς πάνε τα πράγματα. Υπάρχει αυτός ο ανθρωπιστικός αφοπλισμός που ήταν πολύ σημαντικός λόγω του αντικτύπου του στον πληθυσμό και την υποστήριξη των, θεμάτων, θυμάτων στο πλαίσιο του κειμένου της συνθήκης που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Από τότε αυτό θεωρείται καθημερινή δουλειά με τις νεότερες συνθήκες. Ε, ε, τότε όμως δεν ήταν κάτι το δεδομένο πριν αρχίσει να υπάρχει σύμβαση της Σοτάβας. Όπως γνωρίζετε λοιπόν, πολλοί σκοτώνονται από αυτά τα ε, όπλα. Μετά όσοι επιζούν χρειάζονται φροντίδα διαβίου, υποφέρουν από κοινωνικό αποκλεισμό, έχουν ψυχολογικά προβλήματα και βρίσκονται σε οικονομικώς μειονεκτική θέση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η επιστροφή των εκτοπιστέντων, ε, η ανοικοδόμηση καθυστερεί, η οικονομική ανάπτυξη πλήτεται, αποτρέπονται οι επενδύσεις και αυξάνεται το κοινωνικό κόστος. Το φορτίο των, ε, που, που, που υπάρχει για τα κράτη-μέλη είναι πάρα πολύ μεγάλο, για τα κράτη που έχουν άρκες είναι πολύ μεγάλο. Και όλα αυτά είχαμε στο μυαλό μας όταν αποφασίσαμε να υπάρξει αυτή η σύμβαση το 1997. Άλλωστε υπάρχει και στο ε, προήμιο θέλουμε να σταματήσει αυτό ε, ε, αυτός ο πόνος από τις ε, νάρκες κατά προσωπικού και αυτό αναφέρεται και στις βασικές δεσμεύσεις, δηλαδή να σταματήσει η κατασκευή και η προμήθεια ναρκών, η καταστροφή των ναρκών κατά προσωπικού και των αποθηκών, των αποθεμάτων του χρόνου θα έχουν περάσει 20 χρόνια από την έναρξη ισχύω της σύμβασης και πολλά έχουμε να γιορτάσουμε αυτή η σύμβαση θεωρείται μια εξαιρετική συνθήκη αφοπλισμού. 164 συμβαλόμενα μέρη σήμερα έχουν συνεισφέρει στις, ε, στην αποναρκοθέτηση έχει σταματήσει σε αυτά ε, η κατασκευή ναρκών έχουν καταστραφεί 151 εκατομμύρια νάρκες που δεν θα χρησιμοποιηθούν ούτε θα τοποθετηθούν στο έδαφος. Δεν υπάρχει λαθρεμπόριο, ακόμη και σε χώρες που δεν έχουν συμβαλόμενα μέρη, 33 κράτη, ακόμη και αυτά τα κράτη σέβονται αυτό αυτές τις απαγορεύσεις έχουν δημιουργήσει ε, μορατόρια, έχουν ε, αναστείλει την ε, χρήση και παραγωγή τους. Όσον αφορά την αποναρκοθέτηση υπάρχουν 30 από τα 61 που λένε ότι έχουν πληγεί από νάρκες κατά προσωπικού, έχουν ολοκληρώσει την αποναρκοθέτηση. Αυτό σημαίνει εκατοντάδες εκατομμύρια γης που έχουν επιστραφεί για παραγωγική χρήση στους πληθυσμούς και πάρα πολλά άλλα κράτη ολοκληρώνουν αυτή τη στιγμή τη δουλειά τους. Με αυτή την αποναρκοθέτηση, την εκπαίδευση για τους κινδύνους και τη γνώση στην κοινότητα, ο αριθμός των ε, ανθρώπων που έχουν χάσουν τη ζωή τους έχει μειωθεί δραματικά από τη δεκαετία του 90. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ στο να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει παροχή βοήθειας στα θύματα, δηλαδή πώς μπορούμε να τα εντάξουμε ε, στην εθνική πολιτική, τα άτομα με αναπηρίες, στην υγεία, στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στη μείωση της φτώχειας. Έχουμε λοιπόν κάνει πολλά. Έχουμε καταφέρει πολλά. Είναι πολύ εύκολο μερικές φορές να πούμε ότι η απειλή των αρκών κατά προσωπικού είναι υποέλεγχο. Δεν πρέπει όμως να αφήσουμε αυτή την επιτυχία να μας τυφλώσει, γιατί εξακολουθεί να υπάρχει απειλή από την αυξανόμενη χρήση από μη κρατικού φορείς όπλων ε, και αυτό εξακολουθεί να παραμένει ε, μία απειλή σε κάποιες χώρες και πρέπει να εξακολουθήσουμε να επιμένουμε για την οικουμενικοποίηση της σύμβασης. Αυτή η πρόκληση είναι κατεπίγουσα, πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτήν πάρα πολύ ε, σύντομα Βλέπετε εδώ μερικές χώρες, 33 τον αριθμό που είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της ε, σύμβασης. Ε, τα συμβαλόμενα κράτη θέλουν να συντονίσουν ε, τις προσπάθειές τους για οικουμενικοποίηση της σύμβασης. Η χρήση των αρκών κατά προσωπικού είναι περιορισμένη, όμως υπάρχουν κάποιοι ισχυρισμοί, και ισχυρισμοί κρατών που δεν είναι συμβαλόμενα μέρη, που έχουν μεγάλο απόθεμα ε, τέτοιων ναρκών. κάτι που σημαίνει ότι 29 κράτη που έχουν αναφέρει ότι είναι υπεύθυνα ε, για πολλούς επιζώντες, ε, πρέπει να ε, υποστηριχθούν ε, με διάφορα είδη υποστήριξης και ενίσχυσης, ε, ώστε αυτοί οι άνθρωποι ε, που θα, χρησιμοποιήσουν αυτή τη γη μετά κάπως να υποστηριχθούν. Κάτι ακόμη, έχουμε δει την αύξηση του αριθμού των ατόμων που έχουν τραυματιστεί ή σκοτωθεί από τις νάρκες ε, κατά προσωπικού της αυτοσχέδιες από μη κρατικούς φορείς σε διάφορες χώρες το 2007. Ε, το Landmind Monitor είπε 86.000 άτομα 42% ε, είναι παιδιά. Ξέρουμε ότι πολλά, ε, πολλές περιπτώσεις δεν καταγράφονται Ε, παλιά, θυμάμαστε πριν από μία δεκαετία, ήταν 330.000, οπότε πάνω από 500.000 έχουν προσθεθεί. Είναι λοιπόν ε, πάρα πολύ ε, μεγάλα αυτά τα νούμερα. Οι χώρες αυτές που βλέπετε στην οθόνη σας είναι στη διαδικασία εκαθάρισης των ναρκών, έχουν σοβαρά προβλήματα μόλυνσης, αυτές οι χώρες έχουν αναφέρει ότι τα προγράμματα τους ε, δεν ε, έχουν επαρκή χρηματοδότηση, ενώ είναι σταθερό το παγκόσμιο ποσοστό χρηματοδότησης. Πηγαίνει αυτή η χρηματοδότηση στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, επειδή είναι περισσότερα τα θύματα των ναρκών τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι σημαντικό, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ε, χρηματοδοτούνται καλά αυτά τα προγράμματα. Όμως υπάρχουν κάποια κράτη που εφαρμόζουν τη σύμβαση και κάπως ε, ε, δεν παρακολουθούνται, δηλαδή δεν καταγράφεται η δράση τους, όχι γιατί υπάρχουν θύματα ναρκών κατά προσωπικού, αλλά γιατί έχουν μάθει να ζουν με αυτές. Οι κοινότητες ξέρουν ότι είναι νάρκες εκεί, βλέπω ας πούμε, έχουμε δει ότι ας πούμε στη Ζιμπάμπουα, στο σύνορο με τη Μοζαμβίκη, ε, ξυπνούν και προσπαθούν να κάνουν ζιγ-ζαγ μεταξύ των αρκών για να πάνε για παράδειγμα ε, στα, στο σχολείο τους ή να μετακινήσουν τα ζώα τους κλπ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα στη Ζιμπάμπουα και σε άλλες χώρες ε, που ε, τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που στη δική μας γειτονιά δεν θα το ανεχόμασταν, οπότε καλό είναι να μην χάνουμε, να μην ξεχνούμε αυτές τις χώρες. Για να ολοκληρώσω, είναι ένα ζήτημα αφοπλισμού, ένα ζήτημα ανθρωπιστικό, ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ασφάλειας, προστασίας και δημόσιας υγείας. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και να απομακρύνουμε αυτή την απειλή από ε, όλες τις ε, ε, κοινότητες ε, πολύ ε, σύντομα. Το 2025 είναι ένας ε, στόχος πραγματικός. Κάθε χρόνο γίνεται μία παρακολούθηση της πρόοδου μας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η υποστήριξη των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες που είναι αποδέκτες της υποστήριξης και έχει σημαντικό ρόλο για την τήρηση των υποχρεώσεών της και των φιλοδοξιών υπό τη σύμβαση της Γενέβης. Είπαμε ότι η τελευταία αναθεώρηση έγινε στο Μαπούτο της Μοζαμβίκη και είπαν ότι ε, μέχρι το 2025 θα προσπαθήσουν να έχουν ολοκληρώσει τα συμβαλόμενα ε, ε, κράτη τις προσπάθειές τους. Του χρόνου θα πάμε στο Όσλο, θα κάνουμε την αναθεώρηση της σύμβασης, να δούμε τι πρόοδος έχει γίνει γιατί αν υπάρξει η ίδια ενέργεια για να μπορέσει να αρχίσει να ισχύει αυτή η σύμβαση το 1997, θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα πολύ σύντομα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για την ευκαιρία που μου δώσατε, να σας ενημερώσω και με χαρά θα περιμένω ερωτήσεις που ενδεχομένως να έχετε. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω λόγο στην κυρία Τζέιν Κόκκινγκ, διευθύνουσα σύμβουλο στην συμβουλευτική ομάδα για τι Νάρκε. Παρακαλώ, Τζέιν. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι που είμαι εδώ. Είναι τιμή μου να μιλήσω στην επιτροφή σα. Και Εμείς είμαστε ευγνώμονες σε όλους τους ε, συναδέλφους που είναι στην αίθουσα και που έχουν συμβάλει σε αυτή την εκδήλωση. Επίσης, ευχαριστούμε και την Ένωση όχι μόνο ως ένα από τους μεγαλύτερους δωρητές, αλλά ως ένα εταίρος σε ένα αγώνα που αφορά και οργανωτική και πολιτική στόχευσή μας. Να πω επίσης ότι θα σας δείξουμε διάφορες εικόνες κατά διάρκεια της παρουσίασης. Άτομα που διαμένουν στις κοινότητες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και σας ευχαριστούμε που συζητάμε αυτά τα θέματα εδώ θέματα που αφορούν τις ζωές τους. Έχουμε λοιπόν τις εικόνες τους, οι οποίες έστω και ως εικόνες είναι πολύ σημαντικές. Είναι το θέμα που συζητάμε ως παρουσία. Ευχαριστώ. Το 1997 δεχτήκαμε το, λάβαμε το βραβείο Νόμπελ. Πέντε από τα αρχικά μας μέλη ήταν από αυτούς που είχαν κάνει την εκστρατεία για την απαγόρευση των ναρκών που δείξει σε μία συνθήκη για την καταπολέμηση και εξάλληψη των ναρκών. Ο Μαξ Φάντερ είχε κάνει τότε μία διάλεξη στην αποδοχή του βραβείου λέγοντας ότι με την προσπάθειά μας προσπαθήσαμε να αναδείξουμε το μεγάλο πόνο αυτών των ανθρώπων και αυτό ισχύει και σήμερα γιατί η αλήθεια είναι ότι οι νάρκες παραμένουν ενεργές μετά από πολύ καιρό μετά την πάυση των μαχών και σκοτώνουν πολύ περισσότερο από, άλλο, από οποιοδήποτε άλλο όπλο. Έχουμε ένα όπλο δηλαδή το οποίο δεν διαχωρίζει μεταξύ μια γυναίκα που πάει σε ένα πηγάδι για να πάρει νερό, ενό παιδιού που πάει στο σχολείο και ενό μαχητή. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Σήμερα, δύο δεκαετίες μετά τη συνθήκη, πάνω από τα τρία τέταρτα των χωρών παγκοσμίω έχουν υπογράψει τη συνθήκη και θεωρείται σοβαρή παραβίαση του ανθρωπιστικού δικαίου η χρήση ναρκών. Θέλουμε λοιπόν να τελειώσουμε τη δουλειά μας και γι' αυτό πρέπει να θυμάμαστε το ότι έχει πετύχει η συνθήκη αυτή. Perfect. Thank you. Από το 2012 όλες οι χώρες ε, μέλη της συνθήκης είναι μέρη αυτής της συνθήκης που απαγορεύει την αποθήκευση όχι τη χρήση αλλά και την αποθήκευση αυτών των όπλων στην Ένωση. Αυτό συμβαδίζει με, τα, με τις βασικές αξίες της Ένωσης, σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρόθεση της ευεξίας και της, των πολιτών και, το, και της ειρήνης. Αυτές οι αξίες επικοινώνονται από τα τμήματα της συνθήκης όπου η διεθνής κοινότητα δεσμεύεται να καθαρίσει ακριβώς τα αρκοπέδια που έχουν μείνει σε περιοχές που είχαν δει ε, Θα πρέπει λοιπόν να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς να υπάρχει κανένας φόβος. Το 2014 στη διάσκεψη που είχε γίνει για τις νάρκες είχαμε πει ότι θα θέλουμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας μέχρι το 2025. Στο Μαπούτο λοιπόν η επιλογή της οποίας ως πολύ ήταν συμβολική γιατί ε, ένα χρόνο μετά η ίδια η Μοζαμβίκη είχε ανακηρυχθεί τελείως ελεύθερη από νάρκες. Είναι σημαντικό λοιπόν να θυμόμαστε ότι αυτές οι ίδιες χώρες το είχαν πει ότι ο στόχος και η δέσμευση 2025 συμβάλλει στην αναγνώριση της σημασίας του ζητήματος αυτού, ιδιαίτερα οι χώρες οι οποίες είχαν αντιμετωπίσει μακροχρόνιους εμφύλιους πολέμους. Τώρα το 2018 μας λείπουν ακόμα, μας μένουν ακόμα 7 χρόνια και αρκετές χώρες έχουν μείνει πίσω. Ο ΜΑΓ μαζί με το Trust που αφορά χώρες που έχουν μείνει πίσω ξεκίνησαν την εκστρατεία για να την κοινωνία των πολιτών, τη ΜΚΟ και άλλου, ώστε να συλλέξουμε χρηματοδότηση για τι δράσει αυτέ και να διασφαλίσουμε ότι θα προωθηθούν δράσει και θα εφαρμοστούν που θα καταλήξουν στην, ε, στον πλήρη καθαρισμό των αρκών. Δεν είναι οποιαδήποτε εκστρατεία αυτή. Αποβλέπει το να επανενεργοποιήσει ολόκληρο, ένα ολόκληρο τομέα και να προσθέσει στήριξη και βοήθεια που σε όλους αυτούς που θέλουν να κάνουν πραγματικότητα το στόχο 2025. Και μάλιστα ένα άνθρωπο προηγουμένω που χρειάστηκε να φύγει είπε ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Αλλά νομίζω, όπως ήδη υπόθηκε, κατά διάρκεια της εφαρμογής της ε, συνθήκης έγινε πολύ προσπάθεια για την απελευθέρωση των γεών. Και βλέπουμε βεβαίω ότι πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά ώστε να υπάρχει ασφαλής και δημιουργική εργασία ώστε να πετύχουμε το στόχο μας το ταχύτερο δυνατό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη αποτελεί παράδειγμα στην, προς τη διεθνή κοινότητα σε σχέση με τις δράσεις για τις νάρκες. Και πολλές χώρες μας έχουν βοηθήσει. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δωρητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη δράση κατά των ναρκών παγκοσμίω. Και η μισή από τους μεγαλύτερους δωρητές είναι χώρες της Ένωσης. Οι νάρκες και η παρουσία τους αποτελεί επίσης δείκτη καλής διακυβέρνησης και ασφάλειας και ειρήνης σε μια χώρα, γιατί ε, δείχνει και την καλή σχέση μεταξύ κυβέρνησης και πληθυσμού μιας χώρας. Έχουμε τον πολιτικό ρόλο των αντιπροσωπιών στις διάφορες χώρες οι οποίες προσπαθούν να διασφαλίσουν ακριβώς την επίγνωση του προβλήματος στις κοινέ νόμες. Η Ένωση έχει ένα κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσει για την επίτευξη του στόχου του 2025 με την κατάλληλη χρηματοδότηση και την απαραίτητη πολιτική βούληση, αυτός ο στόχος είναι εφικτός για πολλές χώρες. Παρ' όλα αυτά, οι τωρινέ παγκόσμιε τάσει σημαίνουν ότι σε κάποιε περιπτώσει λείπουν κονδύλια. Ευτυχώ αυτό, ευτυχώς αυτό δεν ισχύει σε πολλά μέρη. Η παρατεταμένη σύραξη στην ε, Μέση Ανατολή απέτρεψε την προσοχή της ε, διεθνούς κοινότητας από αυτά τα θέματα. Η νέα ε, κατάσταση ανάγκης για τις νάρκες νομίζω ότι πρέπει να αναγνωριστεί και να α, συνοδευτεί με δράσεις. Είναι σημαντικό αυτό, αλλά είναι επίσης εξίσου σημαντικό να θυμόμαστε ότι αυτή είναι μετάδοση αφορά ελάχιστες χώρες. Οι κοινότητε σε πολλές χώρες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν την κληρονομιά του πολέμου και κάποιες από αυτές μπόρεσαν, μάλλον δεν θα μπορέσουν να ανακάμψει χωρίς διεθνή βοήθεια. Καθημερινά σκοτώνονται γυναίκες και παιδιά από νάρκες και αυτό είναι απαράδεκτο. Η βούληση όμως πολλών χωρών για την επίτευξη του στόχου 2025 νομίζω ότι δεν συμβαδίζει με την διεθνή βοήθεια. Οι νάρκες συνεχίζουν ακόμα να αποτελούν μια πολύ σοβαρή απειλή σε πολλά μέρη και να αποτρέπουν την ανάπτυξη πολλών χωρών. Στη Ζιμπάμπου, ας πούμε, οι αγρότες αρχίζουν να χάνουν ε, ζωικό κεφάλαιο λόγω ακριβώς των ναρκών, το οποίο συμβάλλει στην φτώχεια τους. Στην Καμπότζη υπάρχουν ακόμα ναρκοπαίδια, ένα ναρκοπαίδια για κάθε 54 κατοίκους. Ένα ολόκληρο ναρκοπαίδιο, όχι μια ναρκή, ένα ολόκληρο ναρκοπαίδιο ανά 54 κατοίκους. Πολλές φορές ο κόσμος μπαίνει ακριβώς σε αυτές τις περιοχές ναρκοπαιδίων ακριβώ λόγω οικονομικής ανάγκη. και όπως και στη Βοσνία Ερζεγοβίνη πάρα πολλές ε, περιοχές ακριβώς, σε πάρα πολλές περιοχέ μπαίνει ο κόσμος παρόλο που γνωρίζει ότι υπάρχει σοβαρός κινδυνός από τις συνάρκειες. Για όλε αυτές τις χώρε, λοιπόν ο στόχος 2025 είναι εφικτό. Όμω, αυτό θα γίνει μόνο με πρόσθετη χρηματοδότηση διεθνώς. Θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να κεντρωθούμε και στην ε, συνέχιση της, των ναρκοπαιδείων. Ε, θα πρέπει να πούμε ότι έχει μειωθεί κατά 70% η δυνατότητα ε, καθαρισμού των ναρκοπαιδείων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδότησε τη Ζιμπάμπουε ή την Καμπότζη στην φάση αμέσως μετά την σύραξη και παρά την πρόσφατη προσχώρηση της Τριλάνκα στην ε, συνθήκη, η διεθνής βοήθεια είναι πάρα πολύ χαμηλή προς τη χώρα αυτή. Αμέσως, δηλαδή μόλις έξι μήνες μετά την προσχώρηση της χώρας. Η διεθνής βοήθεια, παρόλο που δεν αποτελεί το μοναδικό κίνητρο, για προσχώρηση είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Οι ανάγκες των ατόμων που επιβιώνουν από τις νάρκες ε, είναι ισόβιες. Η συνθήκη παρέχει, προβλέπει μάλλον επίσης νομικέ υποχρεώσει προ τα θύματα αυτά. Όσο πλησιάζουμε λοιπόν το 25, η Ένωση και οι χώρε μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η βοήθεια προ του επι, θα παραμένει βιώσιμη και σταθερή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την μοναδική συλλογική ευθύνη να βρει υποστηρίξη, να δημιουργήσει υποστηρίξη ώστε να πετύχουμε το στόχο του 25. Όλοι μας θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες τις χώρες μέλη, ώστε να εξαλείψουμε την ε, κληρονομιά αυτών των ναρκοπεδίων στις διάφορες χώρες. Χρειαζόμαστε λοιπόν στη συνεργασία με τα εργαλεία που προλέβονται από το ΠΔΠ 21-27, τα οποία θα μας ε, δώσουν μια θαυμάσια ευκαιρία για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Θα πρέπει να διευρύνουμε ακριβώς και τα θεματικά εργαλεία που αφορούν την εφαρμογή της συνθήκης και αυτό, όπως είπε και ο Χουαν Κάρλος, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό όμως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί όλα αυτά θα πρέπει να συμπληρώνουν και όχι να αντικαθιστούν τη γεωγραφική υποστήριξη, ώστε με τη χρηματοδότηση μετά την, μετά την, μετά την διακήρυξη του το 2014 να μην έχουμε τεράστια κενά. Παραμένει λοιπόν μια, ένα πολύ σημαντικό δυναμικό αλληλοβοήθειας όταν χρησιμοποιούμε διάφορα οικονομικά εργαλεία και χαίρομαι πάρα πολύ που εδώ επίσης μπορούμε να κάνουμε κάτι. Με την επίτευξη των στόχων του 2025 εμείς θα λαμβάνουμε κάτι περισσότερο από μια πολιτική δέσμευση. Θα επιτρέψουμε σε 16 εκατομμύρια άτομα τα οποία καθημερινά ζουν με τον απαράδεκτο κίνδυνο βομβών που δεν έχουν εκραγεί και ναρκών να, να αποφύγουν μια και καλή, να ξεφύγουν μια και καλή από την κληρονομιά του πολέμου. Σας παρακαλώ, βοηθήστε στον αγώνα μας αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Τζέιν. Νομίζω τα μηνύματα όλων των μιλητών μας ήταν πολύ ενδιαφέροντα, αλλά να τονίσω ακριβώς και το πόσο σημαντικό είναι να υπογραμμίσουμε το πώς έχουμε πετύχει λαμβάνοντας υπόψη το τι αντιμετωπίζαμε τη δεκαετία του 90 και τα καταληκτικά σου συμπεράσματα σε σχέση με τις απώλειες χρηματοδότησης και το τι επιπτώσει είχε αυτό, όπως ας πούμε το 75% μείωση των δραστηριοτήτων ε, καθαρισμού σε διάφορες χώρες. Και όλα αυτά σχετίζονται βεβαίω και με αυτά που συζητάμε εδώ στο Κοινοβούλιο για τα οικονομικά εργαλεία και τις δράσεις που αφορούν αυτά τα εργαλεία. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητέ Ο Μάκ ο συναδελφό μας, ε, ζήτησε το λόγο. Θα ήθελα να υποβάλει κάποιες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι αυτές οι ε, δράσεις ε, Ευχαριστώ λοιπόν. Πιστεύω ότι είναι μία από τις ε, πολιτικές μας υποχρεώσεις που όχι μόνο από πολιτική άποψη αλλά και από ηθική είναι έχουν μεγάλη σημασία. Το έργο αυτό πρέπει να γίνει σε αρκετές εμπόλεμες ε, περιοχές ή ε, περιοχές ε, που έχουν περάσει πόλεμο για να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη αλλά και αγροτική ανάπτυξη διότι ιδίω νάρκες απαντώνται σε αγροτικές περιοχές. Ήρθα από μια εκδήλωση με τον Αλεξάνδρα Χουκ ο οποίος συμμετέχει στην αποστολή ε, στην Ανατολική Ουκρανία και μιλήσαμε εκεί για το πόσες ε, νάρκες έχουν τοποθετηθεί εκεί. Ε, δεν είναι κατά προσωπικού αλλά κατά τάγκ. Η Ρωσία δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως καθότι πρόκειται ακόμα για μία ε, διαμάχη που συνεχίζεται. Έχει νόημα να συζητάμε ήδη το πώς θα απομακρυνθούν, ε, διότι θα είναι ένα έργο για μετά τον, ε, τη διαμάχη. Όσον αφορά την Βοσνία Ζεγοβίνη, μιλάμε για άλλα 15 τετραγωνικά χιλιόμετρα τα οποία πρέπει να καθαριστούν Αναφέρατε λόγους, όμως ε, δεν τους κατάλαβα ακριβώς. Είναι ζήτημα χρημάτων, είναι ε, πρόβλημα επειδή δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται. διότι αυτά τα 15 τετραγωνικά χιλιόμετρα θα πρέπει να μπορούμε να τα καθαρίσουμε και επίσης θυμάμαι την δεκαετία του 90 όχι μόνο στην Βοσνία Ζεχοβίνη αλλά και στην Κροατία όταν πηγαίναμε στις περιοχές εκεί, στις εμπόλεμες ζώνες ε, και αρχίζαμε την καθάριση υπήρχαν αρκετές εταιρείε ε, που έκαναν αιτήσει, ε, είχαν αναπτύξει τεχνικές Είχαμε ένα συγκεκριμένο εργαλείο τότε ε, και γνωρίζαμε που έπρεπε να στραφούμε ενώ τώρα τα χρήματα έρχονται από τα μεγάλα μας ε, προγράμματα. Γνωρίζω λοιπόν μια εταιρεία η οποία συμμετείχε. Αν τώρα δήλωνε ότι θέλει να συμμετάσχει, πού θα έπρεπε να απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ποιον θα πήγαινε, για να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Μάικλ ε, και νομίζω ότι αυτή είναι η τελευταία σου ερώτηση και αφορά και εσένα, ε, Φρανκ, όσον αφορά την πρώτη σου ε, παρουσίαση, το ζήτημα της ορατότητας ε, τι γίνεται όταν έχουμε τις απαραίτητες αλλαγές. Και κάτι ακόμα το οποίο θα ήθελα ε, να σημειώσω με βάση τα σχόλια του James ε, την ήπια δύναμη και που ασκούν οι αντιπροσωπείες μας για το έργο το οποίο γίνεται σε αυτές τις χώρες. Αντίστροφα, τώρα, θα ήθελα να σας ζητήσω να κάνετε κάποια τελικά σχόλια, γιατί δεν νομίζω ότι κάποιος άλλος ζητάει το λόγο. Οπότε θα περάσω αρχικά στην Jane Cocking. Ε, θα αφήσω τις ε, ερωτήσεις ε, για τη Βοσνία Ζεχοβίνη και ποιον με ποιον να επικοινωνήσετε στην ε, Επιτροπή. Όμως αρχικά θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω την Επιτροπή που ε, ρίχνει φως σε αυτό το θέμα και μας προσκάλεσε να συμμετάσχουμε, να συμμετάσχουμε σε αυτή τη συζήτηση, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μοναδική στην θέση που έχει ώστε να προσφέρει την ε, ηθική ηγεμονία και την υποστήριξη και την ανάπτυξη δυνατοτήτων σε κυβερνήσεις ε, με περιοχές που έχουν νάρκες. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι ένας ε, μοναδικός συνδυασμός που προσθέτει τρομερή αξία στα όσα μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ε, μπροστά από το επόμενο πι δελτα πι για το οποίο γίνονται ακόμα διαπραγματεύσεις ε, και η περίοδος αυτή είναι πολύ κρίσιμη ιδιαίτερως ε, λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις για το 2025 δεν θα πρέπει λοιπόν να χάσουμε την προσοχή μας από αυτούς τους στόχους ώστε να ενεργοποιήσουμε αρκετές προσπάθειες θα είναι μια σημαντική κίνηση ώστε να επιτύχουμε ε, μια πολύ μεγάλη δέσμευση που έχει γίνει για να μπορέσουμε να την επιτύχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και που και που θα πρέπει να δίνουμε συγχαρητήρια στον εαυτό μας για το έργο που κάνουμε. Χων Κάρλος, τελικά σχόλια. Ε, ευχαριστώ πολύ όλους σας. στο πλαίσιο της ε, σύμβασης των ενδιαφερόμενων μερών ε, ε, σκεφτόμαστε το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στις χώρες για την επίλυση του προβλήματος, το οποίο απαιτεί εσωτερική, εσωτερικό συντονισμό, ώστε το πρόγραμμα να έχει επιτυχημένη ολοκλήρωση. Και αυτό γίνεται στην Βοσνία και είναι κάτι το οποίο προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα σημαντικό ε, πράγμα το να δούμε ε, μια επιτυχία το 2025. Οι εταίροι θα πρέπει να έρθουν να υποστηρίξουν τις κυβερνήσεις τους ώστε να προχωρήσει το πρόγραμμα και αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο της ε, σύμβασης και είναι κάτι το οποίο θα οριμάσει περισσότερο του χρόνου κατά την ε, συνεδρίαση αξιολόγηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ και θα επιστρέψω στους ε, συμμετέχοντες κατατόπους. Η κυρία Αντωνοπούλου, ο κύριος ε, συνταγματάρχης Λιώσνινγκ θα ήθελε να πει κάτι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε θα ήθελα να απαντήσω το ερώτημα για το αν έχουμε λίγα χρήματα. Όχι. Έχουμε λίγη χαμηλή αποδοτικότητα. Για παράδειγμα το 2017 έχουμε ε, δαπανήθηκε το 75% του, ε, του προϋπολογισμού αλλά επετέφθη μόνο το 35% ε, των δραστηριοτήτων που είχαμε προγραμματίσει τουλάχιστον θα έπρεπε να ε, γίνουμε ύποπτοι για όλο αυτό. Έχουμε 800 ε, μικροπεριοχές, ε, έχουμε συγκεκριμένους στόχους, οπότε ο καθένας μπορεί να επιλέξει από αυτό τον κατάλογο που ακριβώς θέλει να εργαστεί Ε, έχουμε δύο μικροπεριοχές. Ε, μπορούμε να ξεκινήσουμε σε μία περιοχή ε, και να ξεκινήσουν σε μια άλλη, πολύ πιο αργότερα από αυτό, η περιοχή δεν κερδίζει κάτι, γιατί ακόμα έχει γύρω τις περιοχές με Επίσης, έχουμε ελλείψεις όσον αφορά το προσωπικό και τις πληροφορίες σε ορισμένε περιοχές. Πιστεύω ότι υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης όσον αφορά την αποδοτικότητα και από τις δύο πλευρές. Από την πλευρά των ε, εθνικών ενδιαφερόμενων μερών υπάρχει μεγάλη αντίσταση όσον αφορά την αλλαγή. Αντίσταση στην ε, ε, προσέγγιση που αφορά την απελευθέρωση γεών ε, και οι δωρητές ε, αργά τώρα υποστηρίζουν την απελευθέρωση γεών. Ε, αυτό αποτε... θέτει προκλήσεις όσον αφορά τις συμβάσεις. Όσοι έχουν εργαστεί με κάτι τέτοιο καταλαβαίνουν τι λέω, οπότε και οι δωρητές θα πρέπει να γίνουν πιο αποδοτικοί η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αργή όσον αφορά την ε, παραχώρηση συμβάσεων. Οπότε και θα πρέπει να το επιταχύνουμε αυτό το θέμα. Θα πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί επίσης. Με τα ε, νέα ταμεία, προενταξιακά ταμεία, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο έγκρισης, προτείνουμε ε, ένα πρόγραμμα που αποκαλούμε ε, κοινότητες ελεύθερες από νάρκες, οπότε μονάχα αυτές θα λαμβάνουν χρηματοδότηση και θα γίνονται πραγματικά κοινότητες ελεύθερες από ε, νάρκες και πιστεύω ότι και άλλες χώρες και άλλες αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλες χώρες θα γίνουν δημιουργικές ούτως ώστε ε, να βρουν ε, τις λύσεις και τις προτάσεις που αναζητούμε όλοι. Ευχαριστώ ε, πολύ. Και τώρα, Φρανκ, πώς ερχόμαστε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο εκδώσαμε το συγκεκριμένο φυλάδιο και στην τελευταία σελίδα σας λέει με ποιον επικοινωνείτε, είναι η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εκάστοτε χώρα, δεν υπάρχει ε, ένας ε, τσάρος της ε, δράσης για τις νάρκες της Βρυξέλλες, όμως άνθρωποι όπως είναι οι Φωτεινοί και ο συνταγματάρχης ε, αποτελούν τα σημεία επαφής ε, στην Βοσνία. Πώς λοιπόν ένας, ένα ενδιαφερόμενο μέρος θα προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έρθει σε επαφή με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην χώρα. Το καλύτερο όμως είναι όταν η κυβέρνηση μιας τέτοιας χώρας έχει ένα σχέδιο με χρονοδιαγράμματα όπου λέει ωραία χρειαζόμαστε δωρητές ε, σε αυτές τις περιοχές ε, για του χρόνου. Ε, στη συνέχεια θα έχουμε αυτές τις εφαρμογές, στη συνέχεια μερικές ΜΚΟ, ιδιωτικές επιχειρήσεις, τάγματα του στρατού. Είναι δική τους λοιπόν ευθύνη να κάνουν βήματα για να εκαθαρίσουν το έδαφος τους από νάρκες. Ευχαριστώ πολύ και αυτό είναι το σημαντικό να έχουμε αυτή την ε, προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω και να συνεργαζόμαστε με τις συμμετέχουσες χώρες. Και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. και χαίρομαι που η Επιτροπή μας έχει τη δυνατότητα να οργανώσει αυτή την ακρόαση και ήταν και πολύ έγκυρη μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. And I am going to do a final plug that there are still some brochures left at the front. Υπάρχουν ακόμα μερικά έντυπα. Ε, μπορείτε να τα πάρετε παρακαλώ. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα επίσης ε, να δώσω την ε, προεδρία στον ε, συνάδελφο κ. Στρατίνα. Good evening, ladies and gentlemen. Let us go uh, to the last. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ας περάσουμε και στο τελευταίο σημείο της ε, ημερήσια διάταξη για σήμερα, το σημείο 8. Την στρατιωτική κοινωτικότητα. Έχουμε την ε, δεύτερη συζήτηση για την ε, γνωμοδότηση της ε, ΣΕΝΤΕ για τη στρατιωτική κινητικότητα. Θα ήθελα να σας πενθυμίσω ότι το χρονοδιαγράμμα για την υποβολή τροπολογιών ήταν στις 12 ε, Σεπτεμβρίου, ήταν, είναι και τις 12 Σεπτεμβρίου 2018. Μέχρι στιγμής είχαμε 127 τροπολογίες και θα ήθελα αρχικά να δώσω το λόγο στον εισηγητή κύριο Κέλαμ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, πρόεδρε, μείναμε μεταξύ μας. Όμως είχαμε μια αρκετά θετική αισιόδοξη πρόεδρε. Έχουν ε, κατατεθεί τροπολογίες από όλες τις ε, ομάδες. Ε, θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για τη συνεισφορά τους. Σήμερα είχαμε μια γνωμοδότηση από τη συνάδελφο Τελίτσκα, οπότε υπάρχει δυνατότητα τώρα να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές κατά την αρχή της εβδομάδας και δεδομένων των ε, τροπολογιών ε, μας προσφέρουν ένα καλό έδαφος ε, για να εργαστούμε για το τελικό κείμενο, διότι ο στόχος είναι να χρησιμοποιήσουμε την διτή φύση όσον αφορά τα δίκτυα μετακίνησης Ε, κάτι το οποίο παρουσιάζεται στην παράγραφο 12 που λέει ότι χαιρετίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ε, για την χρήση των ταμείων που προβλέπονται για, τη, για προγράμματα στρατιωτικής κινητικότητας ούτως ώστε οι οι δομέ να προσαρμοστούν στις ανάγκε τη ε, στρατιωτική ε, κινητικότητας και τα προγράμματα αυτά θα, ε, θα είναι χρήσιμα επίση και για πολιτική χρήση. Θα μπορούσαμε λοιπόν με βάση αυτό να έχουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα διότι η έκθεση αυτή αποτελεί τμήματα της ε, κοινή ε, πολιτικής ασφαλείας και άμυνας και υπάρχει βούληση για την ενίσχυση της ε, στρατιωτικής αυτονομίας της Ευρώπης και ταυτόχρονα να, δημιουργήσουν, να δημιουργήσουμε συνεργίες με το ΝΑΤΟ. Το ένα σημάδι είναι να κρατήσουμε αυτό το momentum και να προχωρήσουμε με το ζήτημα της στρατιωτικής κινητικότητας διότι με βάση τις ε, συνθήκες που γίνονται όλο και πιο πολύπλοκες η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να καθυστερήσει την ε, προετοιμασία της ε, ούτως ώστε να μεταφέρει άμεσα τα στρατεύματά της είτε αυτό αφορά περιοχές ε, συγκρούσεων είτε ε, σε περίπτωση ανθρωπιστικών καταστροφών ή φυσικών καταστροφών αλλά ε, επίσης συχνά ετησίως έχουμε στρατιωτικές ασκήσεις και θα πρέπει λοιπόν να ξεπεράσουμε εμπόδια όσον αφορά τη στρατιωτική κινητικότητα. Ένα άλλο ζήτημα αφορά την νομοθετική εναρμόνιση και την δυνατότητα στρατιωτικών ε, στρατευμάτων ε, ε, να περνούν τα σύνορα των διαφορών κρατών μελών. Είχαμε την επόμενη Τετάρτη την συνάντηση των σκιωδών και είμαστε έτοιμοι ούτω ώστε να γίνει την, τον επόμενο μήνα η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΑΦΕΤ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κέλαμ. Και τώρα μπορώ να δώσω το λόγο στους σκιώδεις. ο κύριος ε, Βάλεν. Ε, θα εκπροσωπήσω όλους τους σκιώδεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κέλαμ ε, για την δουλειά του και θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε τον επόμενο μήνα όλας Ο στρατός μας έχει πρακτική εμπειρία σχετικά με το πόσο δύσκολη είναι η στρατιωτική κινητικότητα και η μεταφορά στρατευμάτων. Και δεν είναι ε, κάτι το οποίο μπορούμε να καθυστερούμε περισσότερο και γι' αυτό θα ήταν καλό να γίνει αυτό το βήμα και να ρίξουμε φως ε, στην κατάσταση. Όσα προτάθηκαν από την Επιτροπή για, την, ε, για το επόμενο ΠΔΠ σίγουρα πήγαμε προς τη σωστή κατεύθυνση και από πλευράς μας το υποστηρίζουμε για να βοηθήσουμε τον, ε, τους στρατούς μας να κινείται πιο εύκολα. Και θα έχουμε ε, αυτήν την ε, στρατιωτική σένκεν όπου άνθρωποι θα μπορούν να μετακινούνται χωρίς γραφειοκρατία και να πρέπει να σταματάνε σε κάθε σύνορα για να συμμετέχουν σε για να συμμετάσχουν σε μια στρατιωτική άσκηση ε, και ε, μετά μπορεί η γραφειοκρατία να μην λειτουργεί ε, καλά. Είναι μια διτή λοιπόν προσέγγιση. Δεν θέλουμε να αφαιρέσουμε μονάχα τα φυσικά και τεχνητά εμπόδια αλλά να υπάρχει και η δικαιοδοσία, ούτω ώστε ο στρατιωτικό πληθυσμό να μετακινείται πιο εύκολα. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για το έργο σα. So, ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, no, no. So, no, no, no, no. I think uh, uh, to discussion is possible only for Η συζήτηση είναι ε, δυνατή μόνο μεταξύ ευρωβουλευτών. Έχουμε κανόνες ε, τους οποίους πρέπει να, να ακολουθούμε ε, και μόνο οι, τα μέλη μπορούν να θέσουν ερωτήματα όμως στη συνέχεια μπορείτε να επικοινωνήσετε. Ε, ε, αν δεν υπάρχει κανένας άλλος να πάρει το λόγο, θα ήθελα να κηρύξω το πέρα στη σημερινή συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας, να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν, να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς και τα μέλη της Γραμματείας. Δέκα η ώρα θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί. Γεια σας.